morning, dear take your seats. We uh, Καλή σας μέρα. Να αρχίσουμε την συνεδρίασή μας. Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση, δηλαδή με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τα ΕΦΗ e e σύνορα. Δεύτερη μέρα της συνάντησης αυτής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις των διάφορων ειδών συνόρων είναι σαφές για όλους μας ότι τα σύνορα διαφέρουν. Ό,τι απόφαση και αν πάρουμε στο τέλος, έτσι κι θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα σημεία διέλευσης. Θα έχουμε τρεις κύριους ομιλητές, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τη δικιά τους άποψη όσον αφορά τα χερσαία σύνορα, τα ενέργεια σύνορα και τα θαλάσσια. Θα ζητήσω από όλους τους ομιλητές να τηρήσουν το χρόνο ομιλίας τους για να μπορέσουμε να έχουμε και αρκετό χρόνο να συζητήσουμε στη συνέχεια. Μετά την ε, παρουσίαση των ε, κύριων αυτών ομιλητών μας θα ζητήσω από τους συναδέρφους να παρέμβουν. Θα μπορούμε να ακούσουμε δύο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά πάλι δύο από τα Εθνικά Κοινοβούλια, έναν Ευρωβουλευτή κλπ. Σας παρακαλώ όσοι θέλετε να παρέμβετε λοιπόν, παρακαλώ να μας ενημερώσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσοι είναι από τα Εθνικά Κοινοβούλια έχετε κάτι έντυπα μπροστά σας που πρέπει να συμπληρώσετε. Έχετε ένα μπλε έντυπο που είναι για το πρώτο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης και το άλλο έντυπο είναι για το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε τον κύριο Μπρόγκουιστ που είναι από την Φιλανδία, ο οποίος θα αναφερθεί στα χερσαία σύνορα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μπλόμκουιστ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε στα χερσαία σύνορα της χώρας μας και πώς πιστεύουμε ότι το πακέτο αυτό για τα φύση σύνορα θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο μέλλον. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για τα 1.300 χιλιόμετρα χερσαίων σύνορων χωρίζονται σε τρία τμήματα. Το πρώτο είναι αυξανόμενες ροές μετακίνησης. Το εξετάσαμε και χθε. Το δεύτερο είναι το προφίλ των ταξιδιωτών και ο τρόπος με τον οποίο μετακινούνται με ιδιωτικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, πούλμαν κτλ. Και το τρίτο είναι οι καιρικέ συνθήκες. Οι ταξιδιωτικέ ώρες έχουν αυξηθεί 20% κάθε χρόνο, όπως βλέπετε από τη διαφάνεια αυτή. Με εξαίρεση το 2014 ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε τις πιο αυξηνόμενες ταξιδιωτικές ε, ροές. Και την τελευταία χρονιά είχαμε μείωση. Το βλέπετε αυτό δεξιά-δεξιά. Θα έχουμε και πάλι αύξηση. Όταν βελτιωθεί η κατάσταση, ο λόγος που υπήρχε μείωση ήταν τα προβλήματα στη Ρωσία σε ένα μεγάλο βαθμό. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε και πάλι αύξηση όμως. Στα ανατολικά μας σύνορα λοιπόν η κατάσταση είναι αρκετά παράδοξη. Συνήθως έχουμε Ευρωπαίους πολίτες και άλλους που θέλουν να υποφεληθούν από την ελεύθερη διακίνηση. Όμως, στα σύνορά μας, 80% των διελεύσεων γίνονται από Ρώσους κυρίως. στα χερσαία σύνορα. Οι πολίτες τρίτων χωρών βέβαια χρειάζονται πολύ προσπάθεια και χρόνο. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε νέα εργαλεία για να διευκολύνουμε τις διελεύσεις αυτές. Έχουμε αυξήσει τις υποδομές μας για να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ροές. Έχουμε αυξήσει λοιπόν τα σημεία διέλευση επίση, αλλά στο μέλλον δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν είναι εφικτό γιατί ο χώρο που έχουμε στη διάθεσή μα είναι περιορισμένο και δεν γίνεται. Επιπλέον όταν μιλάμε για χερσαία σύνορα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι οδικές αρτηρίες είναι συγκεκριμένες και πρέπει να συνεχίσονται και από την άλλη πλευρά, από τη Ρωσία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν λοιπόν οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα, δεν μπορούμε από μόνοι μας. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο την τεχνολογία για να βελτιωθεί η κατάσταση. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε το σύστημα εισόδων-εξόδων. Κάποιος 36 φορές πέρασε τα σύνορα σε λιγότερο από τρεις μήνες και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αν δίνουμε ε, εύκολη διέλευση σε αυτούς που συχνά περνούν ε, τα σύνορα, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε ένα βελτιωμένο σύστημα. Ο συνεροφύλακας μπορεί από ένα τέτοιο σύστημα να δει ότι έχει περάσει πολλές φορές στα σύνορα το συγκεκριμένο άτομα, ότι έχει τηρήσει τον νόμο πάντα και τις διατάξεις, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ένας ε, ταξιδιώτες χωρίς πρόβλημα. Και άλλες αρχές έχουν πρόσβαση σε ένα τέτοιο σύστημα εισόδων-εξόδων όμως στη Φιλανδία. Εδώ βλέπετε ένα διαβατήριο ενός ατόμου που περνάει τακτικά τα σύνορα. Ε, είναι γεμάτο σφραγίδες το διαβατήριο όπως βλέπετε και χρειάζονται 20 λεπτά περίπου για έναν συναριοφύλακα να υπολογίσει πόσο χρόνο έχει μείνει στη χώρα το συγκεκριμένο άτομο. Το εθνικό μας σύστημα εισόδων-εξόδων λοιπόν μπορεί να μας βοηθήσει για το συγκεκριμένο άτομο. Μπορεί να μπει ε, στην Φιλανδία από ένα συγκεκριμένο σημείο διέλευσης αλλά να βγει από κάποιο άλλο. Εκεί δυσκολεύονται κάπως τα πράγματα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι Ρώσοι μπαίνουν συνήθως το πρωί στη Φιλανδία και βγαίνουν το βράδυ. Γι' αυτό και έχουμε δύο στιγμές τη μέρα που οι ουρές είναι μεγάλες στα σύνορα. Αυτή η εικόνα σας δείχνει τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε το χειμώνα με τις κακές καιρικέ συνθήκες. Μπορεί να έχουμε μείον 30 βαθμούς το χειμώνα. Η διάρκεια της ημέρας όπου έχουμε φως είναι πολύ μικρή. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται επίση και ειδικό εξοπλισμό και ειδικέ διαδικασίε σε τέτοιε καιρικέ συνθήκε. Οι διαδικασίε πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο απλέ. Κατά του ε, ελέγχου, τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε πρέπει να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα γιατί όπως είπαμε ο χρόνος και ο χώρος που έχουμε στη διάθεσή μας για τους ελέγχους know, Όπως γνωρίζετε Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε ότι βλέπουμε μάλλον την ισορροπία πώς ε, έχουν οι διάφοροι παράγοντες ανάμεσα στο σύστημα εισόδων-εξόδων και της καταχώρησης ταξιδιωτών. Αν πάντως το νέο σύστημα δεν λάβει χώρα στο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αναγκαστεί η κάθε χώρα από μόνη της να αναπτύξει τέτοια συστήματα, όπως κάναμε και εμείς νωρίτερα. Χρειαζόμαστε ένα κεντρικό σύστημα που να συνδυάζεται και με το ευρωπαϊκό ΛΙΖΑ. Με τη βοήθεια του πακέτου ΕΦΗ σύνορα μπορούμε να βελτιώσουμε τα ταξιδιωτικές ροές και στο μέλλον, χωρίς να μειωθεί ασφάλεια. Γιατί το σύστημα διευκολύνει το έργο των συνοριοφυλάκων. Υπολογίζει αυτόματα το χρόνο που έχει περάσει κανείς μέσα ε, στην περιοχή Σέγγεν. Μπορεί να ταυτιστεί στα σύνορα ένα άτομο και ακόμα κι αν ε, το ταξιδιωτικό του έγγραφο έχει καταστραφεί χαθεί μερικές φορές μπορεί να έχει έξι διαφορετικά διαβατήρια ένα άτομο. Μερικά από αυτά εντελώς νόμιμα να έχουν εκδοθεί. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι λοιπόν να εντοπιστεί ένα τέτοιο άτομο. Επίσης συχνά συμβαίνει να έχει καταστραφεί, να έχει χαθεί ένα ταξιδιωτικό εγγραφό. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουν οι να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Για τους κατοχυρημένους ταξιδιώτες Τώρα, εδώ χρειάζονται δύο λεπτά μόνο για να περάσουν τα σύνορα. Κάτι το οποίο βοηθάει πολύ. Πολλοί σκέφτονται ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα περιορίζεται στον αυτοματισμό. Όχι. Διευκολύνει και τους ε, πραγματικούς φυσικούς ελέγχους. Για κάποιους καταχωρημένους ταξιδιώτες η έλεγχη είναι αυτοματοποιημένη. Στην Φιλανδία έχουμε ήδη κάνει προσωμείωση των ε, αυτοματοποιημένων ελέγχων ε, υπηκών τρίτων χωρών στα σύνορά μας. Οι δικές μας εμπειρίες πάντως είναι πολλά υποσχόμενες. Στο μέλλον θα συνεχίσουμε με το δοκιμαστικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με το Ιουλίζα. E Εν κατακλείδη, θέλω να σας πω ότι από πλευρά της Φιλανδίας το χρειαζόμαστε το πακέτο αυτό εφή σύνορα. Έχουμε καταφέρει με το δοκιμαστικό αυτό πρόγραμμα με ασφάλεια και ικανοποιητικά να ελέγξουμε τις ταξιδιωτικές ροές. Και ακόμα και αν αυτές αυξηθούν, πιστεύουμε ότι με ένα τέτοιο σύστημα θα καταφέρουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βρόνχης. Θα περάσουμε στις αερομεταφορές. Ο Ολλανδός εκπρόσωπος εκπρόσωπος της ε, Ολλανδικής χωροφυλακής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας αγαπητοί εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των κρατών μελών. Εμείς είμαστε η μεθοριακή φορά θα έλεγα στην Ολλανδία και ασχολούμεθα και με το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Συμμετέχουμε στην πιλωτική φάση του προγράμματος για τα ΕΦΗ e e σύνορα είναι υπεύθυνη η Ολλανδική χωροφυλακή για το πρόγραμμα αυτό και ελπίζω μέσα σε 10 λεπτά να σας μιλήσω για την χωροφυλακή αυτή και να σας δείξω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις προθέσεις που έχουμε μπροστά μας στο μέλλον. Πρώτον, στόχος μας στο ΣΥΠΧΟΛ, στο αεροδρόμιο, είναι ο εξής. Εμείς με ολοκληρωμένο τρόπο καλύπτουμε τις ανάγκες φύλαξης του αεροδρομίου του Άμστερνταμ. Είμαστε η αστυνομική δύναμη, η μεθοριακή δύναμη και η δύναμη ασφάλειας του αεροδρομίου. Στην ουσία συγκεντρώνουμε όλες τις αρμοδιότητες και τις αποστολές της αστυνόμευσης του αεροδρομίου. Έχουμε 600 με 700 ε, ε, μεθοριοφύλακες οι οποίοι εργάζονται συστηματικά στο αεροδρόμιο. Πέρυσι είχαμε 55 εκατομμύρια επιβάτες στο Σκύπχολ. Μεγαλώνει συνεχώς σε καθημερινή βάση το αεροδρόμιο αυτό. Όχι μόνο αυτό το αεροδρόμιο αλλά το συγκεκριμένο μας απασχολεί τώρα. Οι ίδιες τάσεις αφορούν και στα αεροδρόμια των δυτικών χωρών, τα περισσότερα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 40% όλων των επιβατών χρησιμοποιούν το αεροδρόμιό μας σαν αεροδρόμιο διαμετακόμισης. στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ έχουμε 65.000 εργαζομένους συνολικά, άμεσα ή έμεσα. Και γενικά προσφέρει το αεροδρόμιο Σκύπχολ γύρω στα 26 δις ε, έχει προσφέρει στον Ολλανδικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν αρκετά αεροδρόμια που ε, διαχειρίζονται άνω του 1 εκατομμυρίου επιβατών σε εβδομαδία βάση στην Ευρώπη μεταξύ των οποίων και το δικό μας. Το θέμα της κινητικότητας λοιπόν είναι σημαντικό για το αεροδρόμιο, είναι σημαντικό για τον επιβάτη και εμείς επειδή είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο των συνόρων είναι ε, φυσικά σημαντικό και για μας σαν σώμα φύλαξης. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην κινητικότητα από τη μία και την ασφάλεια από την άλλη. Έχουμε λοιπόν αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Πώς εμείς θα κάνουμε τους ελέγχους καλύτερα, με ευφιέστερο τρόπο, ταχύτερα, με, το ίδιο, με τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων αλλά και μέσα στους ίδιους χώρους γιατί δεν έχουμε δυνατότητα ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε περισσότερους χώρους. Εν τω μεταξύ αυξάνεται ο αριθμός των επιβατών, από 55 εκατομμύρια θα φτάσουμε στα 70. Απαιτούνται λοιπόν καλύτερες τεχνολογίες και απαιτείται καλύτερη χρήση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. Αυτή ήταν μια μικρή εισαγωγή. Στα επόμενα πέντε λεπτά θα σας δείξω τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει τον τελευταίο καιρό και κάποιες πρώτες ιδέες. Καταρχάς στο ΣΥΠΧΟΛ έχουμε αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου. Έχουμε 36 πύλες ηλεκτρονικού τύπου και θα διευρυνθούν σε 72 μέσα στον επόμενο χρόνο. Εκεί ελέγχεται ε, το γνήσιο των ταξιδιωτικών εγγράφων, ελέγχεται το όνομα του επιβάτη, το σύστημα βασίζεται στην οπτική αναγνώριση, στην αναγνώριση προσώπου και όλα αυτά λειτουργούν στα πλαίσια ε, του μηχανισμού της Ολλανδικής χωροφυλακής. Καλύπτουμε μόνο τις χώρες Σέγγεν ε, και τα διαβατήρια τα οποία έχουν ηλεκτρονική φυσικά πλακέτα. Νομίζω ότι επειδή είναι πρόσφατο το σύστημα δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία σύγκρισης, αλλά οι ηλεκτρονικές πύλες καλύπτουν μόνο το 3% των αναγκών πρέπει να συνηθίσουν και οι επιβάτες στο νέο σύστημα, πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς οι συνοριοφύλακες. Πέρυσι πάντως μπορούμε να πούμε ότι το 18% των επιβατών που πέρασαν από τον ηλεκτρονικό έλεγχο χρειάστηκαν επιπλέον βοήθεια, το 18%. Επίσης χρησιμοποιούμε ε, το πρόγραμμα καταγεγραμμένων επιβατών ήδη από το 2001 αν κάποιος ζητήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα RT, εμείς σαν χωροφυλακή θα κάνουμε ένα πρώτο έλεγχο και εφόσον μπει στο πρόγραμμα τότε θεωρείται καταγεγραμμένος. Απορρίπτουμε κάποιες από τις αιτήσει ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε. Το πρόγραμμά μας περνά από φυσικούς ελέγχους και τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον συγκεκριμένο επιβάτη δίδονται ε, σε μία μικρή κάρτα στον επιβάτη και δεν σωρεύονται, δεν αποθηκεύονται κάπου αλλού. Και αυτό ε, γίνεται επίσης και στα πλαίσια διμερών συμφωνιών όπως ανάμεσα στην Ολλανδία και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύει εδώ και 14 χρόνια και βλέπουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε συλλέξει επίσης και με το EU Επίσης χρησιμοποιούμε και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό θέλει χρόνο βέβαια. Από πλευράς ε, της Ολλανδικής χωροφυλακής μπορούμε να πούμε ότι η καταγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων απαιτεί χρόνο. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από το σύστημα VIS, But we also saw that the implementation of the FIS system was very complex. We had a lot of technical issues. The learning curve of our border guards, well... Λοιπόν, η, ο τρόπος με τον οποίο ασχολούνται, ασχολήθηκαν με τις αλλαγές τα μέλη της Ολλανδικής χωροφυλακής ήταν χρονοβόρος Έχουμε πολλαπλά συστήματα θα έλεγα ε, για τον έλεγχο του επιβάτη και όταν προστίθενται συστήματα επιπλέον αυτό αποτελεί μια επιβάρυνση. Αυτό το οποίο απαιτείται από εδώ και πέρα είναι συστήματα τα οποία μπορεί να αναλάβουν ε, απλές ε, αποστολές όπως το σκάνινγκ έλεγχος του διαβατηρίου. και μέσω της εισαγωγής εφιών τεχνολογιών σίγουρα ο ελεγκτής μπορεί να συγκεντρώσει καλύτερα την προσοχή του στον ελεγχόμενο. Είναι απαραίτητο επίσης να υπάρξουν καινοτόμες λύσεις, ευφυείς καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της κινητικότητας και φυσικά εδώ το βασικό στοιχείο είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση. Όχι μόνο το να έχει κανείς τις πληροφορίες αλλά το να τις χρησιμοποιεί σωστά είναι το θέμα. Αν κάποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες με αυξημένο τρόπο σημαίνει ότι θα πρέπει να συνδυάζει σωστά τα προγράμματα. Και τέλος πρέπει να διασφαλίσουμε ακριβώς την διαλειτουργικότητα των προγραμμάτων, όχι του VIS ή του SIS, όπως επίσης όμως και του προγράμματος για τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία έχουν κλαπεί Όλα αυτά καλό θα ήταν να μπορούσαν να συνδυαστούν μεταξύ τους σε ένα πρόγραμμα, αυτό θα μας έκανε τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χάρσμα. Και πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, για τη συνεδρία αυτή θα καλέσω τους συναδέλφους και από τα Εθνικά Κοινοβούλια να κάνουν τις ερωτήσεις τους, να ζητήσουν χρόνο ομιλίας για να γίνει επικοδομητική η συζήτηση στο τέλος. Καλό τώρα τον κύριο Μπαρσελόριον από την Ισπανία να μας μιλήσει για τα θαλάσσια σύνορα. Παρακαλώ. Ε, Καλημέρα. Στα ισπανικά θα σας μιλήσω εγώ. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είναι βέβαια μια πρόκληση για μένα αυτό. Αρχίζει η παρουσίασή μου. Λοιπόν, είμαι από το 2003 μέλος της αστυνομίας στην ε, χώρα μου. Είμαι αστυνομική αρχή και συνεργαζόμαστε με τους σενάριοφύλακες. Θα σας δείξω ένα μικρό βίντεο με μία επιχείρηση που έλαβε χώρα το καλοκαίρι. Κάπου όπου είχαμε πολλά επεισόδια και συμβάντα. Το βίντεο αυτό ονομάζεται επιχείρηση Μινέρβα και συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι. Έχετε και το βίντεο μαζί με την παρουσίαση μου PowerPoint. Δεν δουλεύει. Τέλος πάντων, το βίντεο συνοψίζει λίγο πολύ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν ελέγχουμε τα σύνορα. Σε ένα λιμάνι έχει πιο μεγάλη σημασία ακόμα. Τι γίνεται με το βίντεο. Να περιμένουμε ένα-δύο λεπτά, μήπως τα καταφέρουμε.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 την δουλειά της αστυνομίας επιτόπου στους ελέγχους. Ωραία, ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια τότε παρακαλώ.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 Okay. It's with music, but okay. It's, Να, ένα μικρό παράδειγμα του πώς γίνονται οι έλεγχοι και στο κάτω-κάτω όχι μόνο στην Ισπανία, σε πάρα πολλές χώρες. Ξέρουμε ότι συμβαίνει το και έρχονται και από άλλες χώρες να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν ένα χεράκι είναι ένα παράδειγμα το τι γίνεται στα σύνορα όλο το χρόνο. Το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, αυξάνεται ο αριθμός ε, των ε, ατόμων που περνάνε τα σύνορα. Εδώ είναι στη Ταρίφα και στη Θέουτα. Uno de los problemas que nos enfrentamos en frontera es que eh, tenemos flujo de... Μπορεί ξαφνικά να έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ατόμων το καλοκαίρι. Τον υπόλοιπο χρόνο θα έλεγα ότι είναι λίγο πολύ ο ρυθμός διέλευσης σταθερός. Το καλοκαίρι όμως όχι. Και έχουμε και πολλές περιπτώσεις, δεν είναι μόνο οι απλοί ταξιδιώτες. Αυτά ήταν ένα μικρό βίντεο, ένα μικρό παράδειγμα για να ξέρετε τι συμβαίνει στα σύνορα. Ωραία, αφού τελείωσε το βίντεο, ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Να περάσαμε στην επόμενη διαφάνεια που δείχνει τους λειτουργικούς στόχους της Μινέρβα όλο το καλοκαίρι. Δεν θέλω βέβαια να μακρηγορήσω εδώ, Το καλοκαίρι είναι η κατάσταση εδώ. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε την γύρω περιοχή κοντά στην Αφρική δηλαδή, τη σχέση της Αφρικής με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. ότι η Αφρικανική Ήπειρος με την Ευρωπαϊκή βρίσκονται τόσο κοντά, αυτό σημαίνει ότι το σημείο αυτό που σας δείχνω είναι σημείο εισόδου πάρα πολλών ατόμων. Την Αλφιφύρα που είναι ε, λιμάνι στην ε, Μεσόγειο και φορτία μπαίνουν στην Ευρώπη από εκεί και φυσικά πολλοί ταξιδιώτες και πολλοί αποτρίτες χώρες. Και βέβαια και διάφορα κουρασγερόπλοι, έτσι. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε την απόσταση ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία. Εδώ και δύο χρόνια είμαι εγώ στα σύνορα και βλέπω ότι έχει υπάρξει μεγάλη βελτίωση της υποδομής, της τεχνολογικής, στην πληροφόρηση. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Οι φωτογραφίες αυτές είναι την Κυριακή που μας πέρασε. Επόμενη διαφάνεια. Να και ο εξοπλισμός. Ήταν λίγο επανάσταση για μας, ε, πρέπει να πω. Παλιά, ε, όλα αυτά γινόντουσαν με το χέρι. Τώρα γίνονται με τα μηχανήματα. Φαίνεται σουρελιστικό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό για μας. Ήμασταν πολύ τυχεροί που μπορέσαμε να έχουμε αυτόν τον εξοπλισμό, ενώ παλιά έπρεπε με το χέρι να βάλουμε τα ονόματα, να ελέξουμε διάφορες βάσεις δεδομένων. Τώρα αυτός ο έλεγχος γίνεται μέσω του ΣΥΣ, της Interpol. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Να, τι βλέπει η αστυνομία στα σύνορα όταν έχει ένα διαβατήριο. Το βάζει στο σύστημα εισόδων-εξόδων και έχει αμέσως τον χρόνο που πέρασε το άτομο στην Ισπανία. Έτσι, πολύ πιο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ε, δεν χρειάζεται να βάζουμε τις φραγίδες όπως έδειξε και ο συνάδελφος πριν σε μία σελίδα διαβατηρίου 8 σφραγίδες. Χρειαζόμαστε πολύ χρόνο αν είναι να τα κάνουμε όλα αυτά με το χέρι. Εδώ είναι ένα παράδειγμα για να δείτε τι βλέπουμε. Μια μικρή έρευνα που κάνει η αστυνομία στα σύνορα με το άτομο όσο εξετάζεται το διαβατήριο μπορεί να ρωτήσει κάποια πράγματα. Και το σύστημα θα απαντήσει αν υπάρχουν κάποιες απάτες ή κάτι άλλο σχετικά με το άτομο αυτό. Εδώ, στις υπέρυθρες και περιόδεις, έχουμε ένα βασικό στοιχείο ασφάλειας. μπορούμε να ξέρουμε έτσι αν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Και αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, τότε μπορούμε να πάρουμε δακτυλικά αποτυπώματα και έτσι να μην έχουμε πια αμφιβολία. Έτσι ξέρουμε κατά πόσο το διαβατήριο ανήκει πράγματι στο συγκεκριμένο άτομο ή όχι. Εδώ βλέπετε τις δράσεις μας στα σύνορα. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι στο λιμάνι βέβαια, να πω πιο σωστά έτσι, όχι στα σύνορα γενικά, στα λιμάνια. Δεν έρχεται πολλοί κόσμος να ζητήσει άσυλο βέβαια στο λιμάνι. Όλο αυτό το καιρό μόνο δύο αιτήσει έχουμε. Τα τεχνολογικά στοιχεία που έχουν μας βοηθούν να πάμε πιο γρήγορα, να τα 150 οχήματα που βλέπετε εδώ που βρέθηκαν ενώ είχαν κλαπεί. Να ένα παράδειγμα, τι μπορεί να δούμε στα σύνορα. Ε, ακριβά αυτοκίνητα δηλαδή που έχουν κλαπεί και εδώ παράνομα λαφρεμπόριο. Όλα αυτά τα συναντάμε. Δεν κάνουμε δηλαδή μόνο έλεγχο διαβατηρίων, έχουμε και όλα αυτά τα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Αυτή η φωτογραφία τι δείχνει. Είναι κάποιοι που φεύγουν με γεμάτες αποσκευές. Δεν νόμιζε κανείς ότι πρόκειται μόνο για καρέκλες και τέτοια πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα μέσα σε αυτό το φορτηγάκι βρήκαμε αυτά. Αριστερά είναι μάλιστα ένας υπολογιστή που είχε κλαπεί από κάποιον ευρωβουλευτή και τον βρήκαμε. Όλα αυτά βρισκόντουσαν μέσα σε αυτό το φορτηγάκι που έφευγε από την Ισπανία για το Μαρόκο. Να, και εδώ άλλα πράγματα. Ό,τι μπορεί να πέρασε από το μυαλό σας ε, βλέπουμε στα σύνορα. Και εδώ χρήματα. Και εδώ κάποιες στατιστικές για το τι κάνουμε στην Αλταμύρα στο, στα σύνορα, στο λιμάνι. Ελπίζω να μην ε, σας έκανα να βαρεθείτε. Απλώς να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή και κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά οτιδήποτε βελτιώνει τη δουλειά μας ακόμα περισσότερο είναι ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. you very much, Mr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαρθελό Αρχώνα. Ξεκινάμε τη συζήτηση τώρα. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών και μετά στους ε, εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Λιθουανικής Βουλής. Σας ευχαριστώ πολύ. Χτες άκουσα με έκπληξη αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι από την Ιταλία. Πράγματι υπάρχει το θέμα της υπέρβασης ε, του ε, επιτρεπομένου χρόνου ε, παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας στόχος το να ελέγχουμε το χρόνο αυτό. Βέβαια ο Κροάτης εκπρόσωπος ρώτησε αν το θέμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις τουριστικές δραστηριότητες. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς Ρώσους οι οποίοι έρχονται στην Λιθουανία για διασκέδαση. Το ίδιο κάνουν και με τη Φιλανδία και αυτό μπορεί να κρατήσει εβδομάδες ακόμα και μήνες. Πρέπει να βεβαιωθούμε λοιπόν ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στους, στον τουρισμό. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε διάφορους τομείς και δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε την κατάσταση. Τώρα, να μιλήσω λίγο για το σύστημα εισόδου-εξόδου της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης. Οι Σουηδοί συνάδελφοι επέμειναν στη λογική των ασφαλών ε, τρόπων ελέγχου των συνόρων. Πρέπει λοιπόν η ασφάλεια να συνοδεύεται από την ευφυΐα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος. Όταν ένας πολίτης τρίτης χώρας μπαίνει ε, στη ζώνη Σέγγεν, ε, πράγματι θα πρέπει να γνωρίζει το τι θα συμβεί από εκεί και πέρα. Ο κώδικας για το Σέγγεν προβλέπει ότι θα πρέπει να δηλώνεται ε, μία διεύθυνση παραμονής. αλλά δεν εφαρμόζεται η απέτηση αυτή από όλα τα κράτη-μέλη. Από τη δική μου εφαρμόζεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστήσει την ανάγκη αυτή υποχρεωτική. Ευχαριστώ. εκπρόσωπος της Ισπανικής Γερουσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και χθες πρωί και απόγευμα τις βασικές προτάσεις για, το για την νομοθετική απόφαση και εγώ νομίζω ότι οι συναντήσεις αυτής είναι ιδιαίτερε διαφωτιστικές για τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Αναγνωρίζω την προσπάθεια λοιπόν ε, η οποία έχει γίνει και την εμπειρογνωμοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα είναι ωφέλιμη για το σύνολο των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Ε, πράγματι η εμπειρία και σαν παράδειγμα των Ολλανδών ε, σύνοριοφυλάκων όπως επίσης για το παράδειγμα της αστυνόμευσης ε, των λιμένων στην Ισπανία βλέπουμε ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να διευκολύνουμε τις διαδικασίες ελέγχου και την ελεύθερη διακίνηση. Αν και ακούστηκαν κάποιες ανησυχίες γιατί ακούστηκε ότι αν ληφθούν τέτοιου είδους μέτρα, είναι μέτρα τα οποία μπορεί να θίξουν ε, τον τουρισμό. Γνωρίζετε ότι η Ισπανία είναι μία από τις χώρες η οποία δέχεται τους περισσότερους τουρίστες ε, στον κόσμο και γι' αυτό θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε την ανησυχία αυτή. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των ε, επισκεπτών αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειώσουμε την σημασία που έχει ο παράγων ασφάλεια, ιδιαίτερα στον κόσμο που ζούμε σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν με τα μέτρα μας να διευκολύνουμε την ελεύθερη διακίνηση και την ε, είσοδο των ε, επισκεπτών με νομοθετικό τρόπο, αλλά από την άλλη θα πρέπει να αυξήσουμε ε, την ε, προσπάθεια για περισσότερη και μεγαλύτερη ασφάλεια. Στα πλαίσια βέβαια στα οποία αναφερθήκαμε χθε. <clears throat> Δύο βασικά συμπεράσματα βγάζω από τη συζήτηση αυτή το κοινοβούλιο στην Ισπανία και η κυβερνητική πλειοψηφία στηρίζει την ομοθετική πρόταση και το νομοθετικό πακέτο το οποίο προετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεύτερον με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για τους λόγους με τους οποίους ήδη αναφέρθηκα στο θέμα της ασφάλειας ότι θα πρέπει να δώσουμε τις περισσότερες δυνατές εγγυήσεις έτσι ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας να μπορέσουν να εργαστούν με τον πιο σωστό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία στα πλαίσια της συζήτησης η οποία θα ακολουθήσει τις, τους επόμενους ε, ε, μήνες ε, να υπάρχει πάντα επαφή με τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Η κυρία Φαγιών. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Θέλω να επισημάνω ότι είναι σαφές, το γνωρίζουμε όλοι, ότι θα υπάρξουν στο επόμενο διάστημα όλο και περισσότερες αφήξεις ε, υπηκών τρίτων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε τα σύνορα και πιο ασφαλή ε, και πιο απρόσκοπτες όλες τις διαδικασίες, πιο ταχύες τις διαδικασίες. Υπάρχουν βέβαια ιδιαιτερότητες που αναφέρατε και εσείς, σε παραδείγματα θερινή περίοδος, χειμερινή περίοδος κτλ. Ε, θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε πιο τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα με τις ερωτήσεις μου, μια και έχετε τη σχετική εμπειρία. Εσείς από τη Φινλανδία μας είπατε ότι έχετε συστήματα διαφορετικά που μπορεί να επιταχύνουν τις διαδικασίες χωρίς να αρκούν ακόμη. Ωστόσο δεν κάνατε καμία αναφορά στο, στην αρχή η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα που κατακρατείτε. Και για πόσο καιρό. Και ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό να μου απαντήσετε. Ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα και τι θα συνιστούσατε σε σχέση με τις βιομετρικές πληροφορίες. Φαντάζομαι ότι θα έχετε εμπειρία και εσείς από τις κάτω χώρες. Μας είπατε ότι στο αεροδρόμιο θεωρείται χρήσιμη, πολύτιμη, την οπτική εικόνα του προσώπου. τώρα λοιπόν που συζητούμε αν Υπάρχει λόγος να κατακρατούνται τα 10 δακτυλικά αποτυπώματα, το ε, οπτικό αποτύπωμα του προσώπου και τα δύο ε, συνδυασμός και όλα αυτά. Θα ήθελα τις δικές σας ιδέες και ταυτόχρονα με μέλημα να μην έχουμε και να μην δίνουμε την εντύπωση ότι έχουμε υπερβολική διακράτηση δεδομένων. Επίσης για τους ε, καταχωρημένους ταξιδιώτες μας λέτε ότι εάν απορρίψετε την ε, εισαγωγή, την καταχώρηση κάποιων στο σύστημα αυτό των καταχωρημένων ταξιδιωτών, η απόρριψη δεν αιτιολογείται. Δεν υπάρχει ένα σύστημα όμως με βάση το οποίο λαμβάνετε τις αποφάσεις σας. Αυτό θα ήθελα να ξέρω και θα το χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον αυτό, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Για δε την τεχνολογία. Η τεχνολογία που εισάγεται είναι πραγματικά τόσο αποτελεσματική ώστε να αιτιολογείται η δαπάνη που θα χρειαστεί. Γιατί αυτό θα βαρύνει ιδιαίτερα στις ε, ε, σκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν τι μπορούμε να επιτρέψουμε, τι μπορούμε να απαγορέψουμε και στη τελευταία ανάλυση πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να μετατρέπεται σε πιθανό ύποπτο ο κάθε ταξιδιώτης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούικαν τώρα, κάτω χώρες και κάτω βουλή. Excuse me. <coughs> Good morning. Κυρία Κέλκεν, είναι το όνομά μου. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το προφέρετε. Ξεκινώντας θα ήθελα να σας πω ε, σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου κυρία Πρόεδρε για την ε, διοργάνωση αυτής της πολύ σημαντική συνεδρίασης. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ τις κατοχώρες αυτών των ευφυών συνόρων. Το κόστος φυσικά θα έχει βαρύνοντα ρόλο. Και ασφαλώς μας ενδιαφέρει πολύ ε, μια συμφωνία σε μια δέσμη για τα ευφύ σύνορα, εφόσον μπορέσει να προχωρήσει. Τρία θέματα θέλω να θίξω σαν προβληματισμό, όχι δηλώσει. προς τον κύριο Χάλσμα των κάτω χωρών. Καλημέρα σα. Καλό όμω και τους συναδέλφου από την Φινλανδία και την Ισπανία να σκεφτούν τι είδου απαντήσει θα μπορούσαν να δώσουν στα ερωτήματα αυτά. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά τον κύριο Χάρσμα, μα λέει ότι θέλει ένα σύστημα με προσώπου και όχι σύστημα εφιών συνόρων με δακτυλικό αποτύπωμα. Δεύτερη ερώτηση. Θα είναι ασφαλές ένα σύστημα με μόνο οπτική αναγνώριση προσώπου. Δεύτερον. Τρίτον. πόσο χρήσιμο θα είναι τον, και πόσο αποτελεσματικό το να αξιοποιηθούν τα στοιχεία αυτού του συστήματος σε δευτερεύοντα, ε, δευτερεύουσα χρήση, την ε, τήρηση του νόμου δηλαδή. Σκοπεύετε να το, ή το έχετε αναλογιστεί αυτό και πόσο χρήσιμο είναι, πόσο αποτελεσματικό. Αυτό το ερωτώ διότι ο καλός συνάδελφος από την ε, Ισπανία, ο κ. Φερνάντες, δεν φάνηκε τόσο σίγουρος ότι είναι χρήσιμο για την επιβολή του νόμου το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε που πρόφερα λάθος το όνομά σας. Ο κύριος Κρίμη από τη Γερουσία της Ιταλίας. <clears throat> Να πω στον Λιθουανό συνάδελφο ότι θα συμφωνήσω με ένα FES σύστημα ελέγχου στα σύνορα. Όμως οι στόχοι τους οποίους ε, έχουμε θέσει, οι σχετικοί με την ασφάλεια, ίσως να ήταν λίγο δυσανάλογα υψηλή σε σχέση με το πραγματικό σύστημα ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι ξεπερνούν τον επιτρεπόμενο χρόνο παραμονής. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις που θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο στρατηγός Χάρσμα, ο οποίος μας μίλησε για ένα σύστημα στα πλαίσια του οποίου οι πληροφορίες για τον επιβάτη δίδονται ή μάλλον καταχωρούνται σε ένα, σε ένα σημείο το οποίο μπορεί να διατεθεί εφόσον ζητηθεί και στον ίδιο τον επιβάτη, κάτι το οποίο νομίζω μπορεί να καλύψει τις ανησυχίες οι οποίες ακούστηκαν χθε γύρω από το πρόβλημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τώρα για τον Ισπανό ε, συνάδελφο, και γύρω από την εφαρμογή των συστημάτων τα οποία προτείνονται στα πλαίσια του τεστ που έχει ξεκινήσει. Στα πλαίσια των συστημάτων αυτών αναφερόμαστε στο θέμα των βιομετρικών στοιχείων, των δακτυλικών αποτυπωμάτων κτλ. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στα πλαίσια μιας κατάστασης αντίστοιχης με το βίντεο που είδαμε. Υπάρχουν φέρι τα οποία αδειάζουν αυτοκίνητα μέσα στα οποία βρίσκονται επιβάτες. Αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν επιβραδύνει τους ελέγχους. Κανονικά δεν θα πρέπει οι επιβάτες να βγουν από το αυτοκίνητο για να υποστούν τον έλεγχο. Λοιπόν, ε, το σύστημα αυτό, εάν πράγματι έχει κάποια δυνατότητα να ξεφύγει κάποιος από τον έλεγχο, δεν έχει νόημα να υπάρχει. Και, α, συγγνώμη, με συγχωρείτε, μια τελευταία ερώτηση για το πρόγραμμα αναγνώρισης ε, στα πλαίσια αυτών που είπε ο Φιλανδός εκπρόσωπος για τους συχνούς επισκέπτες. Ε, το σύστημα αυτό κοστίζει. Γιατί ξέρετε ότι κάπως έτσι είχε προβλεφθεί το προηγούμενο σύστημα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτό τι κόστος έχει και ποιος καλύπτει το κόστος αυτό. Ο ίδιος ο επιβάτης. Thank ε, Σας ευχαριστώ κύριος Διάστε Μέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Γκάλ. Κάποια σχόλια πριν θέσω ερωτήσεις που νομίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμα για όλους μας. Βασίζονται οι παρατηρήσεις αυτές στις εμπειρίες τις οποίες έχω και εγώ ίδιος και γενικότερα στη χώρα μου. Ακούσαμε ορισμένα παραδείγματα για τα σύνορα στον αέρα σε λιμένες ε, και ε, γενικότερα. Είδαμε τι γίνεται στο Σίπχολ, είδαμε τι συμβαίνει στο Μπαράχας, στη Μαδρίτη. Γνωρίζουμε το θέμα των ε, λιμενικών σημείων περάσματος το από υψηλή πίεση πάρα πολύ συχνά και ακούσαμε και τα παραδείγματα για τον έλεγχο στα σύνορα τα επίγεια ανάμεσα σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ρωσία. Έχουμε επίσης δει τι συμβαίνει στην Φιλανδία Γενικά γνωρίζουμε πολύ καλά με διάφορους τρόπους ε, τις μορφές ελέγχου που επιβάλλει η χώρα αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους συναδέλφους των ε, Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχει η Επιτροπή μας για να μπορέσουμε με συγκεκριμένο τρόπο, με παιδαγωγικό τρόπο να κατανοήσουμε την περιπλοκότητα του νομοθετικού πακέτου χρειάστηκε να επισκεφθούμε αυτού του ε, τύπου της, ε, ε, της, της μονάδες φύλαξης αν θέλετε των σύνορων. Το Σίπχολ σαν παράδειγμα είδαμε πόσο περίπλοκο είμαι και σε κλιματολογικό επίπεδο και σε επίπεδο επιφάνειας και σε σχέση με τις ημερήσιες δραστηριότητες, σε σχέση με τις νυκτερινές δραστηριότητες Είδαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μας έδειξαν προηγουμένως οι φωτογραφίες. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται θα συμπληρώσει την απάντηση την οποία έχει ήδη δώσει ο τελευταίος συνάδελφος που πήρε το λόγο. Στο ΣΥΠΟΛ υπάρχει το θέμα της αναγνώρισης του προσώπου, υπάρχει το θέμα, η μέθοδος μάλλον των δακτυλικών αποτυπωμάτων κτλ. Αλλά στο ΣΥΠΟΛ ο επιβάτης business έχει μια κάρτα στη διάθεσή του ηλεκτρονική, πληρώνει για αυτήν και ξέρετε ότι χρησιμοποιεί την κάρτα αυτή για να κόψει την ουρά ας πούμε και δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι πολύ, δεν υπάρχει καθυστέρηση καθόλου. θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτή η κάρτα και τι κοστίζει στον επιβάτη. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μία παρατήρηση η οποία ίσως να συζητηθεί στα πλαίσια και του επόμενου πάνελ. Ε, με βάση τα προϋπάρχοντα συστήματα και στα πλαίσια της συζήτησης για το νέο νομοθετικό πακέτο θα ήθελα να μάθω ποιες είναι αυτές τις οποίες προτείνονται ε, να, έχουν αυτοί που θα κάνουν τον έλεγχο. Δηλαδή θα είναι στρατιωτικοί, θα είναι αστυνομικοί, θα είναι απλοί επαγγελματίες. Αυτό είναι βασικό για να κατανοήσουμε ακριβώς αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στα πλαίσια της επόμενης φάσης. Το ΣΥΠΧΟΛ είναι σαφές ότι ε, υπάρχει ένας ε, μικρός στρατός ο οποίος απασχολείται, είναι υπάλληλοι στρατιωτικοί εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο. Ε, είδαμε στο ισπανικό παράδειγμα ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τον έλεγχο και την διαμετακόμιση ελέγχουν είναι αστυνομικοί. Λοιπόν, ποιοι θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό στο μέλλον θα αντικαταστήσουμε, θα κάνουμε αλλαγές, θα περάσουμε την επεξεργασία των δεδομένων από το στρατιωτικό προσωπικό στο πολιτικό προσωπικό. Υπάρχουν θέματα εδώ, πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα. Ελπίζω να πάρω κάποιες απαντήσεις για αυτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές γιατί νομίζω ότι οι παρεμβάσεις τους ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Ευχαριστώ κύριε Δίας Και τώρα πάλι στους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αλλά σας παρακαλώ πολύ να περιορίζετε τις τοποθετήσεις σας στα τρία το πολύ λεπτά. Γιατί έχουμε αρκετές ακόμη τοποθετήσεις και πρέπει να αφήσουμε και αρκετό χρόνο στους ομιλητές μας για να σας δώσουν τις απαντήσεις. Από την Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο κύριος Απτάλ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το 2013, το, το Φεβρουάριο, κατατέθηκε η πρώτη πρόταση για τα ευφύ σύνορα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. κύριος στόχος του συστήματος εισόδων-εξόδου ήταν να διευκολυνθούν τα συστήματα εισόδου-εξόδου. Η πρόταση περιλαμβάνει την πρόβλεψη για την καταχώρηση δακτυλικών αποτυπωμάτων και των 10 δακτύλων με στόχο την ε, εξασφάλιση στοιχείων για το σύστημα καταχωρημένων ταξιδιωτών, οι οποίοι θα μπορούν να διέρχονται ευχερέστερα τα σύνορα μέσα από αυτόματες θύρες. για τους ε, μη για τους υπηκόους τρίτων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να διέρχονται τα συστήματα αυτά, κατά την αξιολόγηση αυτού του προγράμματος βλέπουμε ότι μπορεί να προκύψει διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν ασχολούνται με πρόσφυγες και έτονται στο άσυλο λένε ότι έχουν επιφυλάξεις ως προς την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα ενός συστήματος το οποίο θα καταγράφει τα προσωπικά δεδομένα 170 ε, εκατομμυρίων ταξιδιωτών από τρίτες χώρες. Για δε την Τουρκία, η οποία έχει ε, λόγω του εμφυλίου πολέμου στην ε, Συρία υποδεχθεί 1.670.000 πρόσφυγες στο, στην επικράτειά της και αντίστοιχα έχει πάρα πολύ σημαντικό αριθμό διελεύσεων και από τα σύνορα με το Ιράκ, εμείς μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζουμε την ιδέα για μια πρόοδο προς ένα σύστημα ευφυών σύνορων. Ευχαριστώ. Uh, next, uh, from... Ευχαριστώ. Από την Κροατία είναι η επόμενη τοποθέτηση με τον κύριο Κρέγκερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εχθές έγινε πιο γενική συζήτηση. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και εργάζονται στο θέμα αυτό και άρα μπορούν να μας δώσουν τις πρακτικές τους τοποθετήσεις. Έχουν μια πρακτική ε, αντίληψη του ζητήματος των ευφυών συνόρων. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη ότι το όλο πρόβλημα έχει χαρακτήρα οικονομικό και αντικειμενικό. Καταρχάς, κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των διερχομένων και εξερχομένων κατά 5 με 10% χωρίς να είμαστε ε, μέλος του συστήματος Σέγγεν, εμείς στην Κροατία έχουμε ένα πολύ υψηλό αριθμό επισκεπτών και για να μπορούμε να επαληθεύουμε την ταυτότητά τους. Θέλουμε ένα καλό σύστημα πάντα με σεβασμό των, ε, του κράτους δικαίου και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το σύστημα που έχουμε στην Κροατία είναι καλό, μεν. Όμως το ερώτημα είναι πώς μπορεί αυτό να ενσωματωθεί σε ένα πιο περίπλοκο ευρωπαϊκό σύστημα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν με απασχολεί το κόστος που θα συνεπιφέρει κάτι τέτοιο, εσωτερικό, δηλαδή κόστος για το εθνικό σύστημα, το οποίο ήδη είναι υψηλό όλο δε μάλλον εάν χρειαστεί το, το πρόβλημα να το αναγάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να έχουμε ένα σύστημα συνεπές λοιπόν με σεβασμό των άνθρωπων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ε, επισκεπτών σε κάθε επίπεδο, δηλαδή και τόσο πολιτικά όσο και νομικά, κάθε ταξιδιώτη, ε, το ζήτημα περιπλέκεται και έτσι η συζήτηση εδώ νομίζω αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα του ότι θα χρειαστούμε οπωσδήποτε πιο ενοποιημένο, πιο ολοκληρωμένο σε τεχνικούς όρους σύστημα. Κάθε χώρα έχει τις εμπειρίες της. Από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε διάφορες πτυχές της οικονομικής και του οικονομικού και κοινωνικού βίου. Όταν λοιπόν δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, στρατηγικά ολοκληρωμένα συστήματα, χάναμε, δαπανούσαμε πολύ ενέργεια σε συστήματα ασύμβατα μεταξύ τους, προγράμματα και συστήματα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσαν να ενοποιηθούν και να δώσουν ε, την αποτελεσματικότητα σε οικονομικούς ε, και κοινωνικούς όρους που αναμένεται. Αυτό που έχω να πω λοιπόν σήμερα και που έχω υπόψη μου σε σχέση με τα προγράμματα αυτά είναι το ζήτημα της ευελιξίας και του κόστους. Θα χρειαστεί πολύ σύντομα να λάβουμε αποφάσεις για το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα παραδείγματι για τη δοκιμαστική ε, περίοδο το, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το αντικείμενο που θα δοκιμαστεί με το σύστημα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μας απασχολήσει και η χρονική διάσταση, γιατί πολύ γρήγορα θα εμφανιστούν νέες τεχνολογικές εξελίξεις και νέες πιέσεις που θα μας καλούν το ταχύτερο δυνατό να προβούμε σε αποφασιστικές αλλαγές στα σύνορα, διότι βλέπουμε άλλωστε και από το φινλανδικό παράδειγμα ξεκάθαρα, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες δεν ε, αρκεί το προσωπικό φύλαξη των σύνορων. Ενώ υπάρχουν άλλες χρονικές περίοδοι όπου αρκεί και περισσεύει. Δηλαδή παρουσιάζει μια ε, εναλλασσόμενη καμπύλη αυτό το, το φαινόμενο των ροών από τα σύνορα. Άρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα τεχνολογικά επαρκές και αποτελεσματικά οικονομικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει Θα πρέπει να κλείσω τον κατάλογο των τοποθετήσεων. Έχουμε τρει ακόμη από τα εθνικά κοινοβούλια, ε, τρεις ακόμη από το Ευρωπαϊκό και δίνω το λόγο βεβαίω στη συνέχεια και στους ομιλητές. Ο κύριος Χαλαχό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, κύριο Μπλουμκουίστ για τα πολλαπλά διαβατήρια που ίσως δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν με τόση ευχαίρεια αυτοί που τα διαθέτουν αν εισηγόταν ένα σύστημα εισόδων-εξόδων. Εννοείται ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί διαβατήριο που δεν του ανήκει. Ένα. Και δεύτερον, η κατάχρηση αυτή πόσο συχνή είναι. Αυτά τα πολλαπλά διαβατήρια τα διαθέτουν άνθρωποι από μια συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα για δε τα σχόλια που ακούστηκαν στη χθεσινή συζήτηση. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση σχετική με τα, με τα ευφύ σύνορα. Ότι μπορεί να ε, δυσκολέψουν τη διέλευση υπηκόντρων των κρατών ή να μετατρέψουν την Ευρώπη σε φρούριο. Όχι, δεν θα αλλάξουν οι όροι εισόδου-εξόδου. Αλλά χωρίς την τεχνολογική αυτή αναβάθμιση θα έχουμε πολύ περισσότερο η καθυστέρηση και κόστος. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Να κάνω. Από το Βέλγιο. Ο Πρόεδρος Επιτροπής των Εσωτερικών, κύριος Φερμέλιν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι νήσι. Δεν απομονώνονται από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν χώρες από τις οποίες μπορεί κανείς να περάσει με μια σχετική ευκολία παρά την περιπλοκότητα των ελέγχων. Εμείς θέλουμε βιομετρικά συστήματα που να ελέγχουν την ταυτότητα του ταξιδιώτη ε, θέλουμε συστήματα αναγνώρισης προσώπου, θέλουμε συστήματα ε, δακτυλοσκοπικά και γνωρίζουμε και εμπειρίες άλλων χωρών όπως την Ισπανία και την Ολλανδία που στηρίζουν τις προσπάθειές τους στα πλαίσια του συστήματος VIS. Ε, Το Βέλγιο δεν είχε δεχτεί καταρχάς την πρόταση η οποία έγινε αλλά νομίζω ότι τελικά θα στηρίξουμε το πακέτο για τα FEE e σύνορα αφού υπάρξει μια μελέτη σε βάθος σε επίπεδο τεχνικό και αφού δούμε και ελέγξουμε τα αποτελέσματα των πιλωτικών φάσεων εφαρμογής. Αυτό το οποίο τίθεται λοιπόν τώρα σαν πρόβλημα είναι το θέμα της πρόσβασης των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας στα στοιχεία των μεθοριακών ελέγχων. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στα πλαίσια των τρομοκρατικών απειλών. Τίθεται επίσης και το θέμα του κόστους του συστήματος αυτού. Ε, ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλές εκτιμήσεις και από ό,τι βγαίνει το κόστος θα είναι ιδιαίτερος υψηλό και από ό,τι φαίνεται θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Σε πάρα πολλές χώρες αντίθετα τα επόμενα χρόνια όπως και στο Βέλγιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια να γίνουν εξοικονομήσεις ε, ε, δαπανών και είναι δύσκολο να κάνουμε εμείς επενδύσεις για τέτοιου είδους συστήματα. Υπάρχει λοιπόν ένα κάποιο κόστος εδώ το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συγκριθεί το κόστος με τα πλεονεκτήματα, με τα ωφέλη, να δούμε τι κοστίζει το σύστημα αυτό στην Ισπανία και στις κάτω χώρες ε, και να δούμε πόσο αποδοτικό οικονομικά θα είναι ένα τέτοιο σύστημα για να κρίνουμε αν πράγματι ένα τέτοιο σύστημα είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό. Κυρία Αλβάρες. Χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε αυτήν την διακοινοβουλευτική συνάντηση η οποία βρίσκω ότι έχει σημασία. Θα ήθελα να σκεφτούμε την δυνατότητα τα κοινοβούλια των κρατών μελών ε, να αναπαράγουν αυτού του είδους τις συζητήσεις στα δικά τους κοινοβούλια είναι κάτι το οποίο δεν έχει ίσως συζητηθεί σε βάθος όπως θα έπρεπε τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς, α, εκτιμώ ότι υπάρχει ένας κοινός στόχος αλλά υπάρχουν δύο βασικές ε, εκφράσεις θα έλεγα για την επίτευξή του. Όσοι καταρχάς πήραν τον λόγο θεωρούν ότι το θέμα των εξωτερικών συνόρων είναι ένα κοινό θέμα, ένα κοινό πρόβλημα και συμπίπτουμε νομίζω όλοι λέγοντας επίσης ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών ελέγχων. Ε, είναι και αυτός ένας επίσης κοινός στόχος. Από ό,τι φαίνεται τώρα, με έμεσο τρόπο υπάρχει μια τάση η οποία λέει ότι ε, διαφοροποιείται εν μέρη, εν πάση περιπτώσει από κάποιες άλλες ε, απόψεις. Ακούστηκαν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με την δυνατότητα να μην υπάρχουν επαρκείς εγγυήσει έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των προσωπικών δικαιωμάτων σε σχέση με τον έλεγχο της αυτότητας, η ανεξέλεγκτη επίσης χρήση των βιομετρικών στοιχείων είναι θέματα τα οποία είναι φυσιολογικό ε, να ε, δημιουργούν ανησυχίες στους βουλευτές. Ποια είναι τώρα η υπόθεση επί της ουσίας. Μπορεί να φαίνεται ότι αυτό που ονομάζουμε εδώ δευτερεύον στόχος να είναι τελικά ο κύριος στόχος. Αν τυχόν είναι έτσι, τότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με πρόβλημα. Πιστεύω πάντως ότι το να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τις εγγύησεις αυτές, στις οποίες αναφέρθηκαν πάρα πολλοί βουλευτές εδώ, δεν πρέπει να το εκλαμβάνετε σαν αντίθεση στην εφαρμογή αυτού του συστήματος. Όμως, αν περιοριστούμε να συζητάμε μόνο τεχνικά και οικονομικά και αφήνουμε σε δεύτερο επίπεδο τα θέματα που έχουν να κάνουν με εργαλεία τα οποία να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών, καταλαβαίνετε ότι κάνουμε μεγάλο σφάλμα. Μεταξύ άλλων, γιατί οι, οι θέσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνονται οι αποστάσεις ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν την ε, ασφάλεια και εκείνους που θέλουν να προχωρήσουμε στο σύστημα. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Η απόσταση να μικραίνει και όχι να μεγαλώνει. Θα ήθελα ο Ισπανός εκπρόσωπος να μας πει ποιος είναι ο μέσος όρος ο χρόνου αναμονής για κάποιον ο οποίος περνά τα σύνορα στο λιμάνι στο οποίο ο ίδιος δουλεύει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ, Κίνγκα. Και εγώ θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με αυτά που ακούγονται για ένα στοιχείο του χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης που έχει να κάνει με την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σύστημα αυτό ΕΦΗ e σύνορα. Είναι κάτι που συζητάμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες Και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτήν την αντίθεση κατά κάποιο τρόπο που διαπιστώνουμε ανάμεσα στις εθνικές εμπειρίες και των εξωτερικών συνόρων τόσο στα αεροδρόμια όσο και στα λιμάνια. Πρόσεξα όλος ιδιαίτερο, τόσα μας είπε ο εκπρόσωπος από το λιμάνι της Αλχεσχύρας που μπορεί να μην το ξέρουν όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι στρατηγική σημασία στο λιμάνι αυτό, πολύ βασικό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτία αν μη τι άλλο του τεράστιου όγκου ταξιδιωτών που τακτικά μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί. Πάνε και έρχονται πολύ συχνά από το Μαρόκο, οι εποχιακοί εργαζόμενοι για παράδειγμα που έρχονται ξανά και ξανά και περνούν από το λιμάνι αυτό. Αυτή ακριβώ είναι η τακτική μετανάστευση που συναντάμε και γι' αυτό και θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι κατάλληλες. Το ερώτημα είναι, έχουμε υπολογίσει τον αντίκτυπο της εφαρμογής του πακέτου αυτού ευθύ σύνορα στη δικιά σας περίπτωση. Ο στόχος σας είναι ακριβώς να διευκολύνετε μέσω αυτού του Μητρώου καταχώρησης ταξιδιωτών, να διευκολύνετε το πέρασμα, τη διέλευση εκείνων οι οποίοι είναι νόμιμοι, τηρούν τους κανόνες κλπ. Πρόκειται για ξένους επισκέπτες λοιπόν που μας έρχονται από το λιμάνι αυτό. Πρόκειται για Μαροκινούς ή άλλους Αφρικανούς. Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος λοιπόν, κατά πόσο θα διευκόλυνε αυτό την πρόσβαση των ατόμων που τηρούν τους κανόνες. Όλο το τοπίο για ενίους κανόνες για τα εξωτερικά σύνορα μερικές φορές έχουν σαν αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται όσοι θα επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν δυνητικά παράνομοι εγκληματίες, κακοί τέλο πάντων. Στιγματίζονται. Υπερβάλλουμε δηλαδή μερικές φορές σε αυτή την αλυσίδα παράτυπης μετανάστευσης που τελικά πρόκειται για θύματα των ε, παράνομων κυκλωμάτων μεταφοράς μεταναστών. Πρόεδρος, από το Εθνικά Κοινοβούλιο, τελευταίο είναι ο κύριος Τότ από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, παρακαλώ, κύριε Τότ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να σας καλωσορίσω εξ ονόματος και και του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Καταγραφής θα ήθελα να πω ότι συνεισφέρει αρκετά στην ε, ε, αίσθηση ασφάλειας στην περιοχή, στην χώρα μου η αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Έχει μεγάλη σημασία σήμερα να υπάρχει πρόσβαση στα συστήματα καταγραφής και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται για να καταπολεμηθεί ε, το η συνοριακή ή διασυνοριακή ε, εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υποχρεωτικά ε, θα επιμηκύνει τους χρόνους αναμονής. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Νομίζω ότι οι σφραγίδες στα διαβατήρια είναι κάτι το οποίο δίδει πληροφορίες όχι μόνο στους αστυνομικούς που κάνουν τον έλεγχο αλλά και στους ε, ίδιους τους επιβάτες. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο ε, μπορεί να βοηθήσει ε, την ε, κινητικότητα των ταξιδιωτών. Όταν εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα και δεν υπάρχουν πλέον σφαγίδες στο διαβατήριο θα πρέπει να βρεθεί ε, μια νέα λύση έτσι ώστε μέσω του ίντερνετ σαν παράδειγμα οι επιβάτες να μπορούν να γνωρίζουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς. Ευχαριστώ. Μας εξηγήσατε λεπτομερώς τους τρόπους ελέγχου ε, των επιβατών στο αεροδρόμιο του Σίπχολ στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Ελέγχου Εισόδων-Εξόδων. Είπατε όμως ότι το 18% που χρησιμοποίησαν τις ηλεκτρονικές θύρες χρειάστηκαν βοήθεια και δεν μιλήσαμε για την άποψη των επιβατών. Το αεροδρόμιο έκανε κάποιες μελέτες στους επιβάτες που πέρασαν από αυτές τις μορφές ελέγχου ε, τι θεωρούν οι επιβάτες, ήταν απλούστερες οι διαδικασίες ελέγχου ή πλέον περίπλοκες και προστατέυθηκαν επαρκώς τα προσωπικά τους δεδομένα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι τώρα. Θα διαθέσω συνολικά 15 λεπτά για απαντήσεις και σχόλια γιατί μας πίεσε ο χρόνος. Με τη σειρά που ακούσαμε τους ομιλητές. Κύριε Μπλόγκβιστ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που απευθύνατε στους ομιλητές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω αυτές που με αφορούν. Ε, συνολικά όμως, χωρίς να αναφέρομαι στους ερωτώντες. Απλώς θα επεκτείνομαι σε κάποια σημεία. Καταρχάς για το Εθνικό Σύστημα Εισόδων-Εξόδων και ποιος διαχειρίζεται τα δεδομένα, για πόσο καιρό διακρατούνται. Θα απαντήσω ότι έχουμε ένα εθνικό σύστημα εισόδων-εξόδων με ψηφιακά δεδομένα, τα οποία διακρατά η συνοριοφυλακή, άρα είναι κάτοχος του Μητρώου, αυτού η συνοριοφυλακή, το οποίο διατηρείται για πέντε χρόνια στη διάθεση της συνοριοφυλακής αστυνομίας και των τελωνίων Άρα και οι τρεις αυτές αρχές έχουν πρόσβαση στα αρχεία εισόδων-εξόδων, μόνο βεβαίως στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Βιομετρικά συστήματα. Και προτίμηση για ε, οπτική αναγνώριση προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα, συνδυασμό και των δύο κτλ. Εμείς αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε περισσότερο την επιλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και γιατί, διότι όλα τα συστήματα που έχουν μέχρι τώρα αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό σύστημα στηρίζονται στη δακτυλοσκόπηση. Έχουμε λοιπόν στα σημεία ε, διόδου τα μηχανήματα, έχουμε την εκπαίδευση ήδη εξασφαλίσει των συνοριοφυλάκων μας και έτσι όταν μιλούμε για ε, πύλες συνόρων που αναφέρουν και οι συναδελφοί από τις κάτω χώρες, αλλά έχουμε και εμείς στο, στα αεροδρόμια μας, ε, χρησιμοποιούμε τη δακτυλοσκόπηση. που θεωρούμε ασφαλές σύστημα. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα το οποίο θα συντονίζει αυτές τις επιλογές μέσα από το EU Υπάρχουν βέβαια θέματα σε σχέση με την καταγραφή προσώπου και αυτό το λέω γιατί, διότι δεν έχουν όλοι οι υπήκοοι των κρατών ε, ε, διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία. Δεν έχει λοιπόν νόημα να καταγράφουμε ε, αποτυπώματα εικόνα προσώπου χωρίς να υπάρχουν τα βιομετρικά διαβατήρια. Δεν υπάρχει αντιστοίχηση. Στα δακτυλικά αποτυπώματα Τίθεται βέβαια ζήτημα για το πόσο διάστημα μπορούμε να κρατήσουμε τα στοιχεία στο σύστημα. Αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την νομοθεσία που αφορά και την πρόσβαση κτλ. αλλά και με τα βιομετρικά στοιχεία και τον αριθμό των βιομετρικών στοιχείων που χρειάζεται να αποθηκεύονται. Εάν λοιπόν έχουμε στο σύστημα εισόδων-εξόδων τα 10 δακτυλικά αποτυπώματα για διακρατούμενα για 6 μόνο μήνες, δυσκολεύουμε για τον ταξιδιώτη την ε, κατάσταση, γιατί θα πρέπει να του πάρουμε και τα 10 δακτυλικά αποτυπώματα μόνο για μια περίοδο 6 μηνών και μετά πρέπει να ξαναρχίσουμε. Άρα η περίοδος διακράτησης δεν εξυπηρετεί μόνο τη συνοριοφυλακή, αλλά και τον ταξιδιώτη, ώστε να αποφεύγονται οι ε, αναμονές στα σύνορα και οι ουρές. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη να το ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος και προχωρήσουμε στην εισαγωγή του συστήματος. Αναφέρθηκε το κόστος από πολλούς ομιλητές και πολλές φορές. Ναι, είναι υψηλό το κόστος της δέσμης ευφυών συνόρων. Το δεχόμαστε, αλλά θέλω να υπογραμμίσω, όπως είχα πει και στην ε, παρέμβαση μου, ότι όπως εμείς, αλλά και η Πορτογαλία, η Ισπανία, κάτω χώρες, έχουμε προχωρήσει ήδη και διαπιστώνουμε ότι θα χρειαστεί να, γίνει, να αναλυφθεί κάποιο μέτρο στα σύνορά μας και ακόμη περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το να εξασφαλίσει ένα σύστημα με μονομενό κράτος μπορεί να σημαίνει δαπάνη εκατομμυρίων, αν όχι δεκάδων εκατομμυρίων. Εάν το κάνουμε όλοι μαζί, ασφαλώς έχουμε οικονομία κλίμακος. Και όπως είπα και στην παρουσίασή μου, Υπάρχουν σημεία εχμής μέσα στην ημέρα, ώρες αιχμής θα έλεγα, όπου φτάνουν μαζικά περισσότεροι ταξιδιώτες και μετά είναι πολύ πιο αραιή η προσέλευση. Έτσι ε, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις ε, διακυμάνεις των ροών. Τα δύο διαβατήρια Τα γνήσια, τα πολλαπλά διαβατήρια που λέγαμε νωρίτερα, είναι γνήσια διαβατήρια. Ε, πολλές φορές βλέπουμε να τα, να τα κρατούν ε, Ρώσοι και υπήκοοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Άρα στα σύνορά μας μπορούμε να έχουμε ανθρώπους και με έξι ή επτά διαβατήρια ακόμα. Μπαίνοντα λοιπόν στη χώρα μπορούν να διαλέξουν ποιο διαβατήριο θα δειξουν στον φρουρό, χωρίς να υπάρχει καμία παρανομία ή παρατυπία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για μας είναι αδύνατον να καταγράψουμε και να παρακολουθήσουμε πόσο διάστημα έχουν μείνει στην περιοχή. Ακόμα και η ορθογραφία των ονομάτων μπορεί να διαφέρει από το Κυργιστάν στο Ουσμπεκιστάν και το καθεξής. Ε, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Κάτι ακόμα που αφορά το κατά πόσο να επιβαρύνεται ο καταχωρημένος ταξιδιώτης με το κόστος. Εμείς ακόμη δεν έχουμε τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό που θα θέλαμε όμως θα ήταν ένα σύστημα ευφυών συνόρων που θα, να ξεκινήσει σύντομα και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε με σύστημα κατηχωρημένων επιβατών. Προς το παρόν έχουμε μόνο σύστημα εισόδων-εξόδων στα εθνικά σύνορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπλόγκβιστ. Ο κύριος Χάρσμα έχει το λόγο. I would like to thank Mr. Diaz de Mera, uh, Mrs. Fayon, uh, but also Mrs. Hallo Allo, who took the, the opportunity to visit Amsterdam Airport. Ευχαριστώ. Καλό θα ήταν ε, να βρεθείτε και να δείτε κι εσείς ποια είναι η κατάσταση επακριβώς που ισχύει στο Σίπολ. Για να έρθω στην ερώτηση της κυρίας Φαγιών. Ρώτησε, είπε αν κάποιος ε, δεν γίνει δεκτός, γιατί δεν ε, ενημερώνεται. Μπορεί να έχουμε βρει κάτι στο σύστημα της αστυνομίας, δεν μοιραζόμαστε την πληροφορία αυτή με καμία άλλη πλευρά όμως. Ούτε με τον ε, εργοδότη, ούτε κανέναν άλλον που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα αρτή. Στο τι μέρα μας είπατε προσοχή σε μια χώρα μπορεί να βρείτε τις αστυνομικές αρχές, σε μια άλλη να είναι στρατιωτική ή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εγώ επίτηδες δεν σας είπα πολλά πάνω σε αυτό, όχι μόνο γιατί δεν είχαμε αρκετό χρόνο, αλλά γιατί ε, περιγράφω τους αυτούς μας σαν ένα είδος χωροφυλακής. Είμαστε δηλαδή μια αστυνομική αρχή με στρατιωτικό καθεστώς όμως. Επίσης ο Δίθεντε Μέρα ρώτησε για το κόστος εισόδου στο πρόγραμμα ΑΡΤΗ. Είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα, πράγματι. Και πρέπει να πληρώνει κανείς συνδρομή ανάλογα με το πακέτο που έχει. Είναι 100 με 200 ευρώ το χρόνο το κόστος για την κάρτα αυτή. Έρχομαι τώρα στην κυρία Κάκεν οι πρώτες δύο ερωτήσεις σας. Τις απαντάω μαζί, αν είμαστε υπέρ ενός πιο απλού συστήματος. Ναι, φυσικά. Όσο πιο απλό, τόσο το καλύτερο. Γιατί θα βοηθήσει την ροή ταξιδιωτών στα σύνορά μας. Συνεπώς, είμαστε σε μια δοκιμαστική περίοδο που αρχίζει τον επόμενο μήνα και θα δούμε τι θα γίνει με την κινητικότητα κατά πόσο όταν κάποιος δίνει μόνο δαχτυλικά αποτυπώματα ή και αναγνώριση προσώπου και θα δούμε κατά πόσο για τα δαχτυλικά αποτυπώματα είναι αρκετά 4-8 ή παραπάνω. Εξοικονομούμε. Λέτε, όχι, αλλά ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα όσο γίνεται πιο απλό σύστημα, που συγχρόνως όμως να μας προσφέρει όσο γίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Για την τρίτη σας ερώτηση, κυρία Κάλκεν, έχει να κάνει με την, τις αρχές επιβολής του νόμου και την πρόσβασή τους, κατά πόσο αυτό είναι το δευτερογενές ή όχι. Αν μπορούν έτσι να είναι πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι, ναι. Αλλά ως συνοριοφίλικες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια πολιτική διάσταση εδώ. Αν συνδέσουμε με το πακέτο ευφύ σύνορα, τις αρχές επιβολής του νόμου. Από πλευρά συνοριοφυλάκων πάντως θα ήμασταν υπέρ του να εισαγάγουμε ένα τέτοιο σύστημα. Για τον κύριο Κρίμη τώρα από την Ιταλία. Ε, ρωτήσατε κατά πόσο αποθηκεύονται τα ταξιδιωτικά στοιχεία. Τουλάχιστον αυτό καταλάβατε. Όχι, εμείς την ταξιδιωτική ιστορία δεν την αποθηκεύουμε. Ναι, θα ήταν, θα μου βοηθούσε. Αν μπορούσαμε να δούμε την ιστορία του ταξιδιώτη που έχει πάει. Δεν αποθηκεύουμε τέτοια ε, στοιχεία ούτε στα πλαίσια του API ε ούτε στα πλαίσια του PNR. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι όταν κοιτάει κάποιος στο διαβατήριο, ε, βλέπει την ταξιδιωτική ιστορία, βλέπει από πού μετακινήθηκε προς τα πού στις τρίτες χώρες, εκεί που χρειάζεται θεώρηση αν μη τι άλλο. Στον κύριο τώρα για το κόστος και το θέλει. Δύσκολο μπορώ εγώ να απαντήσω. Το πρόγραμμά μας RT εδώ και 14 χρόνια ισχύει. Δεν θα μπορούσα όμως να σας δώσω απόλυτη απάντηση. Θα πρέπει όντως να αξιολογηθούν το θέλει και το κόστος και ευχαρίστω αν θέλετε μετά να το συζητήσουμε διμερώς. Να απαντήσω τώρα και στην κυρία Ροβό, κατά πόσο έχουμε ερευνήσει καθόλου με τους επιβάτες πώς εκείνοι βλέπουν την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Το έχουμε κάνει, όχι βέβαια επιστημονικά απόλυτα ικανοποιητικά θα έλεγα, αλλά έχουμε συζητήσει με τους επιβάτες και αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι τους ικανοποιεί. Πρέπει να το συνηθίσουν βέβαια, παρόλο που είναι απλό. Παρ' αυτά είναι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται να γυρίσει στη δεξιά σελίδα του διαβατηρίου. Στην αρχή μπορεί να του δυσκολεύει λίγο, αλλά του ικανοποιεί γενικά και δεν έχουμε ακούσει τίποτα παράπονα όσον αφορά το θέμα της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Χάρσμα. Τελευταίος ο μιλητής, ο κύριος Μπαρθέλο. Bueno, Ευχαριστώ. Πάω επί της ουσίας, Μια που είμαι στην πρώτη γραμμή, όντως έχω πολλές πληροφορίες. Χωρίς όμως να μπορώ να πω ότι τα ξέρω όλα. Για, θέμα, τα, για παράδειγμα το ποιος αποθηκεύει τις πληροφορίες και πώς τις αποθηκεύει, δεν τα ξέρω. Για να απαντήσω στην κύριο Κλήμη για το ΑΜΠΕΣΕ. Πρέπει να σας πω ότι τα συστήματα αυτά εφαρμόστηκαν στην ζώνη των επιβατών. Στα οχήματα δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστεί το σύστημα αυτό. Το λιμάνι μου έτσι είναι πιλωτικό λιμάνι για τέτοιου είδους ελέγχους. Είναι πάντως πάντα θετικό. Οι πύλες αμπεσέ, δηλαδή, η αυτοματοποιημένη συνοριακή έλεγχη, είναι δοκιμαστικό για να δούμε πώς μοιράζεται η ροή ταξιδιωτών από τρίτες χώρες με εκείνους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα τις ροές αυτές. Για τα οχήματα δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Στον κύριο Άλβαρες για το χρόνο αναμονής. Το καλοκαίρι είναι κάτι που δεν εξαρτάται μόνο από την αστυνομία. Εξαρτάται και από τα πλοία. Πόσο γρήγορα αναχωρούν. Για να έχετε μια ιδέα, από τη στιγμή που φτάνει το πλοίο μέχρι που να περάσει, μιλάω για τα οχήματα τώρα, να περάσει από το φίλτρο των σύνορων 45 λεπτά, μισή ώρα. Εξαρτάται. Εξαρτάται και από το τι θα βρούμε. Δηλαδή περνάνε τα οχήματα και εξαρτάται τι θα συναντήσουμε. Τι χαρακτηριστικά θα, έχει το κάθε όχημα και το τι θα βρούμε στο κάθε όχημα. Αλλού πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο για τις ραγίδες, να ελέγξουμε περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν ε, βελτιωμένο, αν υπάρχει αυτοματισμός δηλαδή, αν δεν χρειάζεται εμείς να βάζουμε τα στοιχεία στον υπολογιστή, αλλά αυτόματα το μηχάνημα τα παίρνει και τα ελέγχει, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι κέρδος. Τώρα για τους εποχιακούς εργαζόμενους που έρχονται στην Ισπανία για δουλειά, συνήθως είναι γυναίκες που έρχονται για τη συγκομιδή φράουλας και συνήθως πριν έχουμε τον κατάλογο που πριν έτοιμο. Έπειτα υπάρχει και το VIS που ελέγχει τις θεωρήσεις και μπορούμε τη θεώρηση να τη βάλουμε στο μηχάνημα και εκεί βλέπουμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή, αν έχει αλλάξει κάποια φωτογραφία, συγκρίνουμε πότε την πήρε την θεώρηση και έτσι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Με τη θέωτα δεν ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Γι' αυτό σας λέγω, είμαι στην πρώτη γραμμή, δεν έχω όλες τις πληροφορίες. Για τον κύριο Τίθ Δεμέρα, να του πω τη γνώμη μου, είπε ότι ναι, είμαστε αστυνομικοί, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Και καταρχήν θέλουμε να έχουμε τις πληροφορίες που μας χρειάζονται για τον κάθε άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι είμαι τίμιος. Έχουμε περάσει έτσι κι αλλιώς από πολλά φίλτρα. Έχουμε ελεγχθεί δηλαδή για να αναλάβουμε τη δουλειά αυτή που κάνουμε. Είμαστε αστυνομία, μην το παίρνετε άσχημα. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι δεν είναι έντιμοι και καλοί, αλλά έχουμε ελεγχθεί για να προστατεύσουμε εμείς και τους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και αυτούς οι οποίοι περνούν τα σύνορα. Εγώ δεν συμπεριφέρομαι άσχημα στους ε, μετανάστες ούτε καν σε κάποιον που θα έρθει και θα αποδειχτεί ότι έχει πλαστό διαβατήριο ή αν διαπιστώσουμε ότι έχει κάνει κάποια πάτη, κάποιο έγκλημα. Πολλοί από αυτούς έτσι καλώς τους έχουν ε, ξεγελάσει στις χώρες τους, τους έχουν πουλήσει ένα πλαστό διαβατήριο. Ε, τους λέω, λυπάμαι πολύ, πρέπει να σας γυρίσω πίσω. Δεν είμαστε οι κακοί. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα. Και θέλουμε να έχουμε τα μέσα για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας για να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Αυτά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος της ε, τρίτης ε, στρογγύλης τράπεζας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για, τους παρε... για τις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές. Ήταν πολύ χρήσιμη ε, η συνάντηση μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Θα διακόψουμε λίγο για να αλλάξουν θέσεις ε, τα μέλη του πάνελ. Ο εκπρόσωπος της Πορτογαλικής Βουλής ε, θα έρθει να να προεδρεύσει ο κύριος Μαγκαλιάης και επίσης ο κύριος Σάρων και η κυρία Μπρόμπαρ. Okay, dear colleagues, uh, Συνεχίζουμε, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Μαγκαλιάς. Όλοι γνωρίζετε τη διαδικασία πλέον. Γνωρίζετε ότι το θέμα τώρα είναι πολύ ευαίσθητο, είναι το θέμα των, της πρόσβασης των δυνάμεων ασφαλείας στα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα νέα προγράμματα. Έχουμε δύο μιλητές. Ο ένας θα έρθει πολύ σύντομα, θα δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή και θα έχουμε χρόνο μετά περίπου μία ώρα για συζήτηση. Λοιπόν, από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας θα ακούσουμε την κυρία Σέλενα. τον κύριο Σέλενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να τοποθετηθώ σε σχέση με την καταπολέμηση της νομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ελπίζω να μπορέσω να επεκταθώ και σε διάφορες πτυχές των εφιών συνόρων και να σας προσφέρω τρόπο το την συνδρομή μου τόσο στο οργανωμένο έγκλημα όσο και στην τρομοκρατία κυρίες και κύριοι διαπιστώνουμε διεθνοποίηση αλλά και εξειδίκευση των ε, δραστών. Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκές αργονές που αποτελούν πρόσφορη αγορά για το οργανωμένο έγκλημα και δίνουν δυνατότητες για καταμερισμό εργασίας και επαγγελματική ανάπτυξη. Η διεθνής τρομοκρατία βρίσκει στη Δύση χώρο και για ε, επιστράτευση μελών αλλά και για δράση. Βλέπουμε λοιπόν προπαγάνδα, επάνδρωση, συντονισμό, επικοινωνία των εγκληματικών ομάδων που αναπτύσσεται και στον πλασματικό κόσμο αλλά έχει οπωσδήποτε και φυσική παρουσία αναγκαστικά για τις οργανώσεις αυτές, οι οποίες ε, δεν μπορούν να δρουν αποκλειστικά και μόνο στον πλασματικό, τον εικονικό κόσμο, αλλά πρέπει να έχουν και φυσική σωματική παρασία. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα ταξιδιών, η διακίνηση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις οργανωμένες αυτές εγκληματικές οργανώσεις. Και αυτό καθώς μάλλον αυτές οι οργανώσεις έχουν όλο και πιο υψηλού επαγγελματικού επίπεδου συνομωτική δράση, κατάρτιση, για να αναγνωρίζουν και τα μέτρα της αστυνομίας, για να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, για να συγκαλύπτουν τις επικοινωνίες τους Επίσης μπορεί να καλύπτονται ή να υιοθετούν πλαστά ή κλεμμένα ονόματα και στοιχεία ταυτότητας δραστηριοποιούμενες στους, ε, στο χώρο της Ευρώπης. Σε αυτήν την ε, περίπτωση πάντως πρέπει να στηρίζονται ε, σε, να στηρίζονται σε αξιόπιστους συνεργάτες και χάρη σε αυτούς να μπορούν να αποφεύγουν τον έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών και της αστυνομίας και να είναι βέβαιες ότι αυτοί δεν θα είναι πράκτορες βέβαια της αστυνομίας ή των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε να κάνουμε με ε, οργάνωση που καλύπτει επιμελητία, σχεδιασμό επιχειρήσεων, εξυπηρέτηση στόχων και με τη χρήση υπηκών τρίτων κρατών με ε, παραδείγμα τη συγκαλυμμένους ε, στόχους ταξιδιού, Εμφανίστε κάποιος ως επιχειρηματίας που ταξιδεύει ή μπορεί να χρησιμοποιεί ε, νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν στη θέση τους νόμιμα και γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα στη διάθεση των, ε, των ε, τρομοκρατικών ή εγκληματικών οργανώσεων. Έτσι λοιπόν οι αρχές ασφαλείας των κρατών μελών κάνουν ό,τι μπορούν για να αναγνωρίσουν και να αντιδράσουν εγκαίρως στις ε, επιθέσεις των κλιματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Βλέπουμε ωστόσο ότι πολλές φορές είναι υποχρεωμένες να αντιδρούν μετά τα γεγονότα και αυτό μας το δείχνουν περιπτώσεις όπως ε, επεισόδια και χτυπήματα όπως το Παρίσι, της Βρυξέλλες, στην Κοπενχάγη. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε ωστόσο και στο πλαίσιο των εφιών συνόρων για την ανάγκη εξισορρόπησης της ελευθερίας με την ασφάλεια. Εξισορρόπηση η οποία είναι πολύ σημαντική αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εγώ θα δώσω έμφαση περισσότερο στην ασφάλεια γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Εάν λοιπόν ε, διακίνηση υπηκών τρίτων κρατών σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερη ε, ασφάλεια, περισσότερες συνθήκες ασφαλείας, αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο και μπορώ ακόμη και χωρίς να είχα στη διάθεσή μου την διετή φάση αξιολόγησης που έχουμε αναπτύξει ε, να τοποθετηθώ ε, προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή βλέπω ότι η εμπειρία που έχουμε από τα εθνικά συστήματα, το εθνικό σύστημα εισόδων-εξόδων ε, βελτιώνεται η ασφάλεια χωρίς να επηρεάζεται η ευχέρεια διέλευσης του ε, ταξιδιώτη και αυτό είναι η προσωπική μου διαπίστωση ως ειδικό. Ωστόσο τα συστήματα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν πανάκια τα συστήματα εισόδων-εξόδων. Ε, Μπορούν να δώσουν όμως μια δυνατότητα για να ξεκαθαρίσει το μοσαϊκό σαν εικόνα, να γίνει δηλαδή πιο καθαρή η εικόνα, αλλά και στα επιμέρους σημεία του, στα κομμάτια του δηλαδή το μοσαϊκό αυτό, να ε, μας εξηγήσει πώς χρησιμοποιούνται από τις εγκληματικές ε, οργανώσεις οι δυνατότητες διακίνησης ποια μέτρα, ποια μέσα χρησιμοποιούν για να ε, καταχραστούν τα, ε, των συστημάτων του κράτους δικαίου και της ασφάλειας. Έτσι μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτά, τα, αυτές τις εγκληματικές κινήσεις. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό δηλαδή εργαλείο με το οποίο μπόρεσαν να αποτραπούν αρκετές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε αποτελεσματική δίωξη τρομοκρατικών και εγκληματικών οργανώσεων στην Ευρώπη. Ένα σύστημα εισόδων-εξόδων που σημαίνει επαγγελματικότητα φυσικά και ασφάλεια. Παρουσίασα κάπως αφηρημένα την κατάσταση μέχρι τώρα. Τώρα θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ξεκινώ λοιπόν με τα μέσα για τα οποία έχει γίνει μέχρι τώρα λόγος, έστω και ακροθυγός. Ένα, τα δύο από αυτά μάλλον είναι τα πρώτερα οι πρώτερες πληροφορίες ταυτότητας, API και το PNR, το ε, Μητρό Όνομα των Επιβατών. Εδώ λοιπόν έχουν, έχει χρησιμότητα να δούμε την διαφοροποίηση μεταξύ διελεύσεως ε, χερσαίας ή Βλέπουμε παραδείγματι τους ε, μαχητές οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Συρία όχι μόνο αεροπορικός αλλά και χερσαία διαξηράς. Εκεί τα συστήματα PNR API δεν μας βοηθούν. Το σύστημα πληροφοριών Schengen μπορεί νομίζω να αξιοποιηθεί περισσότερο και να δώσει καλά αποτελέσματα στην περίπτωση των μαχητών, μόνο όμως εάν καταγράφεται κάποιος σε ένα σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και ταυτόχρονα μπορεί στη γραμμή ελέγχου στα σύνορα να εντοπιστεί και αναλόγως βέβαια να ε, υπάρξει σχετική αντιδρασία από τις αρχές. Εάν όμω ε, την ώρα που ταξιδεύει κάποιο δεν έχει μπει στο σύστημα πληροφοριών Schengen, δηλαδή οι πληροφορίε σχετικέ ε, κοινοποιούνται μόνο μετά το ταξίδι του, τότε δεν βοηθάει πολύ το σύστημα SIS. Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα πληροφοριών θεωρηστιβατήριων, VIS. Μπορούμε να κάνουμε επαλήθευση των στοιχείων του ετούντα, αλλά δεν μας ε, λέει το σύστημα αυτό εάν έχει ταξιδέψει προς τη Συρία από τον ευρωπαϊκό χώρο κτλ. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τρίτα κράτη τα οποία δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών θεώρηση διαβατηρίων, το VIS και δεν το χρησιμοποιούν. Καθένα λοιπόν από τα εργαλεία που σας προανέφερα έχει λόγω ύπαρξης και χρησιμότητα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Αλλά να είμαστε και ρεαλιστές, δεν αποτελεί κανένα από αυτά πανάκια και δεν υπάρχει κανένα μέτρο το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική λύση συνολικά σε ένα φαινόμενο ε, το οποίο είναι περίπλοκο. Μόνο συνδυασμός μέτρων και μέσων μπορεί να δώσει αποτελεσματική καταπολέμηση το φαινομένου της τρομοκρατίας. Τώρα, το θέμα των ευφυών συνόρων δεν βλέπω να αλλάζουν πολλά πράγματα, διότι κύριος στόχος καταρχάς είναι η μετανάστευση του συστήματος των ευφυών συνόρων, άρα θεωρώ ότι είμαι ε, μόνο δευτεραγωνιστή στη συζήτηση που γίνεται εδώ, μόνο παρεπιπτόντος μπορεί να αξιοποιηθεί το σύστημα εισόδων-εξόδων, Πιστεύω όμως ότι ένα σύστημα εισόδων-εξόδων παρόλα αυτά παραμένει αξιόλογη βοήθεια για τις αρχές επιβολής του νόμου. Και τους, τις διευκολύνει πολύ στο να αντιδρούν εγκαίρως έναν ενδεχομένο κίνδυνο. Ας δούμε λοιπόν αφενός με τη δίωξη, αλλά στην αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν για να δούμε την αποτροπή κινδύνων. Που σημαίνει τι, ότι θα μπορούμε ταχαίως και κατά τρόπο οργανωμένο, δικτυωμένο να αναλαμβάνουμε δράση. Αυτό θα σήμαινε για τον ειδικό που είμαι τη δυνατότητα χωρίς ιδιαίτερες περιπλοκές και διατυπώσεις να έχω πρόσβαση στην εικόνα του υπόπτου, να έχω μια σαφή εικόνα για τα στοιχεία του και να μπορώ να αντιδρώ σχετικά γρήγορα. Παραδείγματα από το τομέα της διεθνού τρομοκρατίας. Και ξεκινώ με το εξή σενάριο, σημειώνοντας ότι δεν είναι τόσο πλασματικά ή φανταστικά τα σενάρια αυτά που θα σας αναφέρω. Φυσικά σας παρακαλώ να αντιληφθείτε και να δεχτείτε ότι όσο και αν ανάγονται στο παρελθόν οι περιπτώσεις που θα αναφέρω δεν μπορώ να δώσω πραγματικά στοιχεία και ονόματα. Τα έχω κάπως αλλιώσει λοιπόν. Παράδειγμα, η υπηρεσία με την οποία συνεργαζόμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η υπηρεσία λαμβάνει ενημέρωση σήμα ότι κινδυνεύει να εκδηλωθεί τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι καθόλου συνηθιστό. Είναι πολύ συνήθες να λαμβάνουμε τέτοιου είδου πληροφορίες τις οποίες καλούμεθα να ε, αξιοποιήσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε. Λαμβάνει λοιπόν και διαβιβάζει αυτή την πληροφορία. Ε, μας λένε ότι οι ύποπτοι προέρχονται από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Έχουμε κατακαιρματισμένες πληροφορίες από την συνεργαζόμενη αυτή υπηρεσία του τρίτου κράτους. Σε συνεργασία όμως με τα εθνικά λειτουργικά μέσα προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε εκείνους που βρίσκονται στη Γερμανία που θα εντασσόταν στο προφίλ του υπόπτου και επίσης ενημερωνόμαστε ότι ε, έρχεται ως ε, διαχειριστής του σχεδίου επιθέσεως ε, κάποιος εκτός Γερμανίας για το σχεδιασμό και την εκτέλεση. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος έχει προσχεδιάσει, έχει επισκεφθεί τους χώρους επιθέσεως, έχει εντοπίσει και προσελκύσει ε, τους ε, εκτελεστές και τους έχει προετοιμάσει. Έρχεται λοιπόν από το εξωτερικό το άτομο αυτό για να κάνει την εποπτεία στο χώρο, στους χώρους της επιθέσεως. Ξέρουμε συγκεκριμένα για αυτό το άτομο ότι υπάρχουν πέραν των πραγματικών και νόμιμων στοιχείων και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στη διάθεσή του, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία μπορεί να προέρχονται από, ε, από κλεμμένα γνήσια ε, ταξιδιωτικά έγγραφα και συχνά λευκά, ε, παρθένα δηλαδή ταξιδιωτικά έγγραφα γνήσια, όπως συνέβη πολύ συχνά στη Συρία και το ξέρουμε αυτό, ότι έχουν εκλαπεί συχνά γνήσια αλλά παρθένα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία συμπληρώνονται στη συνέχεια. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση στην οποία εμείς χρειάζεται οπωσδήποτε να ξέρουμε αν το άτομο αυτό έχει γνήσια έγγραφα, στη διάθεσή του έχει πλαστή ταυτότητα και αν με αυτά τα γνήσια ή την πλαστή ταυτότητα έχει έρθει, έχει μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε πέραν των στοιχείων που μας δίνει το ε, συνεργαζόμενο το ε, κράτος εταίρος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, με στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι γνήσια, εάν όντως έχει μπει εντωμεταξύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να μας το δώσει το σύστημα μέχρι τώρα. Εάν δεν πρόκειται για κάποιον που ταξιδεύει με πλαστά έγγραφα ή εναλλάσσει ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως άλλωστε εξετέθηκε νωρίτερα, προφανώς δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Η βιομετρική όμως διάσταση εδώ θα μας βοηθούσε πολύ για να αναγνωρίσουμε επαρκή στοιχεία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό εάν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει εξέλθει της χώρας το άτομο αυτό. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει ολοκληρώσει την αποστολή του. Το σχεδιασμό τον έχει ολοκληρώσει και άρα περνάμε σε μια άλλη φάση όπου οι εκτελεστές ενδεχομένως έχουν επιφορτιστεί με, το, με την επίθεση και άρα συγκεκριμενοποιείται περισσότερο ο κίνδυνος για μια τρομοκρατική επίθεση. Εάν έχει πραγματοποιηθεί αυτή η έξοδος από τη χώρα, Άρα έχει αυξηθεί ο τρομοκρατικός κίνδυνος, έχει ενταθεί ο τρομοκρατικός κίνδυνος. Πρέπει εμείς να ενισχύσουμε σημαντικά τα μέσα προστασίας. Άρα πρέπει να ξέρουμε εάν και να ε, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μια σειρά από τα οποία θα μας δώσουν όσο το δυνατόν πιο σαφή εικόνα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι για μας να αναγνωρίζουμε εφόσον έχουμε εντοπίσει μία δομή δικτύου, εάν και άλλα μέλη του δικτύου αυτού έχουν ταξιδέψει προς ή και έξω από τη χώρα, έχουν εξέλθει από τη χώρα. Άρα εδώ θέλουμε να βλέπουμε όχι μεμονωμένα γεγονότα. Θέλουμε όσο δυνατόν, ειδικά όταν πρόκειται για τρομοκρατία, ε, να βλέπουμε και να μπορούμε να διαγνώσουμε αν πρόκειται για παράλληλες πολλαπλές επιθέσεις ε, μεταχρονολογημένες επιθέσεις, διαδοχικές δηλαδή επιθέσεις και άρα θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι είδους κίνηση υπάρχει για τα εμπλεκόμενα στο δίκτυο αυτό άτομα στην χώρα και σε διαφορετικούς ακόμη τόπους και προορισμούς. Αυτά πρέπει να μας τα δίνει το σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό. Στην πραγματικότητα όμως, στον κόσμο που ζούμε, τα στοιχεία αυτά μας, τα, μας φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση. Δεν υπάρχουν προκαταβολικά στη θέση των υπηρεσιών ασφαλείας, μόνο ύστερα από ε, ανάπτυξη δράσεων των διοκτικών αρχών, κατοικών έρευνε, συλλήψεις, ανακρίσεις, μπορούμε να δούμε, εκ των υστέρων υπογραμμίζω, ότι έχουν πραγματοποιήσει τις κινήσεις αυτές εντός και εκτός της χώρας τα εμπλεκόμενα ε, άτομα. Ένας, Απτούλ Αλχασάν, πλαστό όνομα σας δίνω τώρα, ε, βλέπουμε ότι πριν από δύο εβδομάδες μπήκε στην ε, Γερμανία, ε, συνάντησε τρεις δράστες, υποψήφιους δράστες, εκ των οποίων, οι οποίοι επί παραδείγματι είναι Βόρειο Αφρικανοί, τους έδωσε τις οδηγίες τους και στη συνέχεια βγήκε από τη Γερμανία. Εδώ έχουμε να κάνουμε κατακαιρματισμένα στοιχεία, τα οποία όμως πρέπει να είμαστε θέση να συνδυάσουμε για να ε, κάνουμε την ε, ανοικοδόμηση του δικτύου, να, να, να φτάσουμε να αναπλάσουμε το δίκτυο και να καταλάβουμε τι σημαίνει. Η αποθήκευση των στοιχείων τώρα. Η αποθήκευση των στοιχείων έχει μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε και να βαθμολογήσουμε τον κίνδυνο και τον παράγοντα κινδύνου έχουμε σχετικά καλή εμπειρία και πιστεύω ότι στην περαιτέρω συζήτηση μπορούμε να ε, καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη λύση η οποία και να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα, την ανάγκη προσωπικών δεδομένων αλλά και να μας δίνει επαρκή ε, προστασία της ασφάλειας. Κλείνω εδώ το παράδειγμα και το σενάριο που θέλω να σας παρουσιάσω. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ότι έχουμε υπηκόους τρίτων κρατών που φεύγουν από την Ευρώπη για να μπουν ως ενοπλημαχητές στην Συρία. Δηλαδή στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει αυτά τα λεγόμενα κύτταρα ε, τρομοκρατικά κύτταρα, τα οποία όμως διασπούν για να πάνε να πολεμήσουν στη Συρία. Αυτό είναι ενδιαφέρουσα πληροφορία για μας. Και βλέπουμε με αυτό ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου κάποιος έχει εξέλθει της χώρας και μόνο μετά την έξοδό του μπορούμε με ασφάλεια να τον κατατάξουμε ως τρομοκράτη υποψήφιο ή τζιχαντιστή όταν επί εμφανίζεται ε, στο YouTube ως τζιχαντιστής, μέλος του λεγόμενου ε, Ισλαμικού κράτους και τότε μόνο αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε το πρόσωπο αυτό και να συλλέγουμε τις πληροφορίες πότε μπήκε, πότε βγήκε από τη χώρα, να συλλέγουμε τα στοιχεία ε, για την ταυτότητά του και να αναγνωρίζουμε αν πρόκειται για κάποιον ο οποίος ε, μπορεί να θεωρηθεί για την ε, διάπραξη και άλλων τρομοκρατικών δράσεων. Ε, επίσης θα ήθελα να επεκταθώ κλείνοντας σε άλλους χώρους της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα στα ναρκωτικά, έχουμε αντίστοιχη δράση των δικτύων, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν την επιμελητιακή εποπτεία μιας επιχείρησης και ταξιδεύουν εντός και εκτός της χώρας. Εάν εμείς λοιπόν μπορούμε να λάβουμε αυτή την πληροφορία ότι αυτός που έχει την επιμελητική διαχείριση των μεγάλων καρτέλ των ναρκωτικών μπαίνει στη χώρα, στην Ευρώπη ή βγαίνει από την Ευρώπη, συνδυάζοντα την πληροφορία αυτή με άλλα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα, μπορούμε να έχουμε ενδεχομένω την εικόνα για την οργάνωση ενό ευρύτερου ε, λάθρεμπορίου ναρκωτικών. Και βέβαια αυτό σε συνδυασμό και με άλλε δραστηριότητε στο κράτο στόχο. Αυτό συνδυαζόμενο λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε για τις εισόδους, εξόδους, γενικά τη διακίνηση των ατόμων αυτών, που μπορεί να προέρχονται από ένα καρτέλ και που είναι ύποπτα για ε, λαθρεμπόριο των ναρκωτικών. Όπω είπα, συνδυάζουμε εκτό των εσόδων-εξόδων και άλλα στοιχεία που έχουμε στη διαθεσή μα και τότε μπορούμε με πολύ πιο στοχευμένο τρόπο να εντοπίσουμε του υπόπτου και να του ε, ε, αποτρέψουμε με το σύστημα εισόδων και εξόδων συμπληρώνουμε σημαντικά κομμάτια του μεγαλύτερου μοσαϊκού, της ευρύτερης εικόνας, την κάνουμε πιο σαφή την εικόνα αυτή και γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω να μην λησμονηθεί η πτυχή αυτή της ασφάλειας. Γιατί ναι πρέπει να εγγυόμαστε και την ελευθερία στην Ευρώπη, αλλά οπωσδήποτε και την ασφάλεια. Επιτρέψτε μου δε να πω ότι εδώ η κατάσταση που έχουμε δεν είναι είτε είτε. Όταν η κατάσταση της διακινδύνευσης είναι τέτοια, πρέπει να, έχουμε τη, να, δώσουμε τη δυνατότητα της αντίδρασης στις αρχές και αυτό χάρη στην αναγνώριση των σχεδίων ταξιδιού των υπόπτων. Έτσι και ο δικός μας ο κόπος θα ε, περιοριστεί, θα είναι πιο ευχερές το έργο μας, αλλά και θα διευκολύνουμε τη διακίνηση εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι δεν εμπλέκονται στις δραστηριότητε. Γιατί θα μπορούμε πολύ γρήγορα και πολύ στοχευμένα να προχωρούμε στους, στους ελέγχους εκείνους που θα επιτρέπουν την αποτροπή τρομοκρατικών κινδύνων από τις αρχές. Μια και δεν έχω πολύ χρόνο παραμένω και διατελώ στη διάθεσή σας, ε, δεν έθιξα πολλές άλλες πτυχές του, του ζητήματος, αλλά πολύ ευχαρίστως εάν έχετε με τις ερωτήσεις σας ανάγκη για περαιτέρω διευκρινήσεις να απαντήσω και δίνοντας ενδεχομένως περαιτέρω παραδείγματα για να εξηγήσω ποιες είναι οι ανάγκες των αρχών ασφαλείας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα, όσα μα είπατε για τους κινδύνου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Εβελίν Μπράουερ, η οποία διδάσκει, όπως γνωρίζετε, μεταναστευτικό δίκαιο στη νομική σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, Free University Amsterdam. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι τιμή για μένα που με καλέσατε ως ειδικό για τα θέματα αυτά που εξετάζετε σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ τους οργανωτές λοιπόν και θα σας πω ποια είναι η άποψή μου για την προστιθέμενη αξία που έχει το πακέτο FEE ε, σύνορα και η πρόσβαση σε αυτό των αρχών επιβολής των, του νόμου. Εγώ ως ερευνήτρια θα σας μιλήσω αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Μέιερς που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση στο Άμστερνταμ που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Θέλω να τονίσω τρία κριτήρια πρώτα απ' όλα που πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικά σε αυτά που συζητάμε εδώ. Και αυτά είναι η νομιμότητα, η αναλογικότητα και η αποτελεσματικότητα. Αυτά τα τρία κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. Γιατί όπως ξέρουμε και από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, αν δεν λαμβάνονται υπόψη αυτά, τότε καταδικάζονται πράξεις οι οποίες δεν τα τηρούν. Πριν μπω λοιπόν στις λεπτομέρειες, επιτρέψτε μου να σας δώσω δύο παραδείγματα από τη δικιά μου εμπειρία που μου ήρθαν στο μυαλό όταν ε, άκουσα για το θέμα της βάσης δεδομένων και των ελέγχων στα σύνορα. Θυμάμαι από προηγούμενες έρευνες που είχα κάνει την δημιουργία τότε του Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών Σέγγεν, το ΣΥΣ. Πριν από αυτό είχα συναντηθεί με διάφορους αξιωματούχους, βλέπετε και την ηλικία μου, πριν καν αρχίσει να λειτουργεί και θυμάμαι ότι είχαν εκφράσει πάρα πολλές αμφιβολίες για την εφαρμογή ενό τέτοιου συστήματος τόσο ευρεία βάσης δεδομένων δηλαδή. Φοβόντουσαν αυτή την συνεργασία και τις ανταλλαγές απόψεων γενικά σε ένα ευρύ πλαίσιο και προτιμούσαν τις διμερείς σχέσεις και τις διμερείς επαφές με ανθρώπους που γνωρίζαν. Γιατί νιώθαν ότι θα χάναν τον έλεγχο στις υποθέσεις που εκείνοι είχαν αναλάβει αν υπήρχε ένα τέτοιο ευρύ σύστημα βάσης δεδομένων. Σήμερα ξέρουμε ότι θεωρείται πολύ πετυχημένο το ΣΥΣ, ακριβώς εξαιτία των κριτηρίων που περιλαμβάνει. Αυτό λοιπόν μου θυμίζει πάντα πόσο σημαντικό είναι το θέμα της εμπιστοσύνης όταν θέλουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες με άλλες αρχές. Το δεύτερο παράδειγμά μου έχει να κάνει με κάτι που διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε ότι το 1 τέταρτο των αστυνομικών στην Ολλανδία που εμπλέκονται σε έρευνες για εγκλήματα και του ζητήθηκε να δώσουν το DNA τους προκειμένου να αποκλειστούν από τις ευθύνες αρνήθηκαν να το κάνουν είπαν ότι ε, φοβούνταν ότι μπορεί να μπλεκόντουσαν ε, τα δικά τους ε, τα στοιχεία, όπως εξήγησε κάποιος αξιωματούχος, γιατί δεν θέλουν να αποθηκεύονται τα στοιχεία τους αυτά σε μια κεντρική βάση δεδομένων, γιατί φοβούνται ότι μπορεί κάποιος να τα έκλεβε ή να υπήρχε κατάχρηση. Επιμένω λοιπόν στο θέμα της εμπιστοσύνης, γιατί πιστεύω ότι είναι προϋπόθεση για να πετύχει οποιοδήποτε νέο μέτρο στην Ευρώπη. Θέλω τώρα να επικεντρωθώ στο εξή. Τι έχουμε, τι θα έχουμε και τι χρειαζόμαστε, τι χρειαζόμαστε παραπάνω. Πρώτα για το θέμα της αποτελεσματικότητας. Όντως, τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε, αυτό πρέπει να ξέρουμε. Και πρέπει να υπάρχει ένα σαφής ορισμός για τα σύνορα. Πάντως, όταν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν ε, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, συμφωνούμε για τους εξή ε, σκοπούς. Ότι θέλουμε να αποφύγουμε την παράτυπη μετανάστευση, ότι θέλουμε να αποφύγουμε να ζητάει κανείς άσυλο όπου είναι πιο εύκολο να το πάρει και θέλουμε και να διευκολύνουμε την νόμιμη μετανάστευση, την ε, σύμφωνα με τους κανόνες μετανάστευση και την ελεύθερη διακίνηση. Και να αποφύγουμε βέβαια την ε, τρομοκρατία και να έχουμε δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Όταν μιλάμε λοιπόν για την μετανάστευση, ξέρουμε ότι έχουμε το σύστημα VIS και το σύστημα Eurodac, που είναι δηλαδή τα δακτυλικά αποτυπώματα που παίρνουμε σε κάθε άνθρωπο που υποβάλλει αίτημα για άσυλο. Οι βάσεις αυτές είναι προσβάσιμες στις αρχές επιβολής του νόμου. Το λέει η ρύθμιση ΒΑΙΕΣ έτσι κι αλλιώς ρητά και λέει ότι ο κύριος στόχος είναι να αποφύγουμε απειλές στην εσωτερική ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας μέλους. Και από τις 20 Ιουλίου του 2015, φέτος δηλαδή, θα υπάρχει πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου και στο Eurotac. Σημειώστε ότι αυτά τα συστήματα έχουν να κάνουν με υπηκός τρίτων χωρών και την καταχώρησή τους στο VIS και το Eurotac και εν μέρη και στο SIS δεν έχει σχέση με εγκληματικές έρευνες ή υπόνοιες, ή υποψίες. Καθαρά για λόγους μετανάστευσης και πέρα από τη χρήση του SIS για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ή για το σύστημα API, την προθυμένη δηλαδή ενημέρωση για στοιχεία επιβατών, δεν έχουμε ένα ευρύ σύστημα που να συμπεριλαμβάνει και ε, προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Μια κεντρική τέτοια βάση έτσι κι αλλιώς είχε απορριφθεί όταν είχε γίνει συζήτηση για τον κανονισμό όσον αφορά τα βιομετρικά διαβατήρια. Τι χρειαζόμαστε τώρα επιπλέον. Μετά τις δολοφονικές επιθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και πιο πρόσφατα στο Παρίσι και στην Κοπεχάγη, ε, Προφανώ είναι απόλυτα θεμητό να θέλουμε αποτελεσματικά μέτρα για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους επιθέσεις που απειλούν την ασφάλειά μας. Η πολιτική θεωρούν ότι τα εφή σύνορα και το σύστημα PNR πρέπει να είναι ψηλά ψηλά στην ημερήσια διάταξη για να αποφύγουμε ακριβώς τέτοιες απειλές. Συζητώντας όμως αυτά τα μέτρα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τους εαυτούς μας και να πρέπει να αναρωτηθούμε τα στοιχεία που θα έχουμε στο σύστημα εισόδων-εξόδων ή στο PNR θα μας βοηθήσουν πραγματικά να αποφύγουμε τέτοιες ε, απειλές για την ασφαλειά μας. Δεδομένου ότι οι δράστες στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήδη γνωστές στην αστυνομία, τους παρακολουθούσε η αστυνομία και οι αρχές ασφάλειας. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο τι είναι αυτό που δημιούργησε τις επιθέσεις αυτές και τι είναι αυτό που μας εμπόδισε να τις σταματήσουμε. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι είναι πολλές φορές Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν βγει καν ποτέ από τη χώρα τους. Οπότε σε τι θα βοηθήσει η πρόσβαση των ε, αρχών επιβολής του νόμου σε ένα σύστημα εισόδων-εξόδων. Σήμερα η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για την πρόσβαση αυτή των αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης είπε ότι η μελλοντική χρήση ε, θα ληφθεί υπόψη στην τεχνολογική αρχιτεκτονική. Δηλαδή, το ακούσατε και χτες, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και επέκταση της διατήρησης των δεδομένων για πέντε χρόνια. Γιατί οι αρχές επιβολής του νόμου θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερος ο χρόνος ο διατήρησης τους. Είναι πιο χρήσιμο αυτό για τη δουλειά τους. Κατά τη γνώμη μου πάντως η απόφαση πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου και η διάταξη για τεχνικά εργαλεία είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί μόνο εφόσον έχουμε συμφωνήσει προηγουμένως για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των συστημάτων εισόδων-εξόδων και καταχώρησης ταξιδιωτών για λόγους μετανάστευσης ως κύριο σκοπό. Άρα πρέπει να υπάρξει ενδελεχής ανάλυση και να έχουμε και όλες τις ρήτρες ασφαλείας που χρειάζονται, ώστε το σύστημα αυτό να έχει μεγαλύτερη νοημότητα. Το θέμα τώρα της αναλογικότητας απορρέει από την θεμελιώδη αρχή για το δικαίωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ξέρουμε ότι έχουν ληφθεί και σχετικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκείνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8 Απριλίου 2014, μια απόφαση DRI, λέει ακριβώς ότι η διατήρηση δεδομένων, η οδηγία σχετική με τη διατήρηση δεδομένων είναι άκυρη, γιατί ακριβώς αδιακρίτως συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς να τα επεξεργάζεται και χωρίς να συνδέει τη συλλογή αυτή με εγκληματικές έρευνες. Η απόφαση αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πριν να αποφασίσουμε και οθετήσουμε την πρόταση για τα ευφυή e e σύνορα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την απόφαση αυτή του δικαστηρίου αν δεν θέλουμε το μέτρο αυτό να κυρωθεί και πάλι κάποια στιγμή εφόσον κάποιος προσφύγει στο δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν και η απόφαση αυτή τρίτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά και άλλες αντίστοιχες. Και βάσει αυτών υπάρχουν και άλλα θέματα θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων που πρέπει να ληφθούν απόψη πριν υιοθετήσουμε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση. Το θέμα της ελεύθερης διακίνησης, για παράδειγμα της επανένωσης των οικογενειών και της μη διάκρισης. Θα ολοκληρώσω με τρία συμπεράσματα. Πρώτον, η αποτελεσματικότητα σημαίνει ότι πριν υιοθετήσουμε νέα μέτρα πρέπει να αναρωτηθούμε τα εξή και να δώσουμε και απαντήσεις για ποιο στόχο χρειαζόμαστε ποιο εργαλείο. Η ερώτηση αυτή έχει να κάνει και με το πεδίο εφαρμογή του εργαλείου που σκεφτόμαστε να εφαρμόσουμε. Οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν μόνο με μη Ευρωπαίους πολίτες. Τελικά ψάχνουμε ανθρώπους μήπως που έχουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα και που μπορεί να αποτελούν απειλή. Και ποιο είναι αυτός ο οποίο ε, αποτελεσματικά μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να εντοπίσει και να βρει αυτόν που απειλεί την ασφαλειά μας. Δεύτερον, οι αρχέ της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας. Σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε πρέπει να βασίζεται σε ε, πράγματα τα οποία να έχουν να κάνουν με την πολιτική μας, να ξέρουμε δηλαδή τι πολιτική εφαρμόζουμε. Αν λοιπόν ξέρουμε ότι το Eurodac θα ε, αξιολογηθεί το 2018, γιατί να μην περιμένουμε μέχρι τότε. Και γιατί να μην καθίσουμε να κοιτάξουμε τι είναι αυτό το οποίο δεν λειτουργεί καλά στο σύστημα πληροφοριών της Europol, που ισχύει εδώ και τόσο καιρό. Γιατί δεν λειτουργεί και τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε σε αυτό. Πριν αποφασίσουμε λοιπόν για νέα μέτρα, θα έλεγα και οι εθνικοί βουλευτές και οι ευρωβουλευτές να ερευνήσουν στις χώρες τους ποια είναι τα κενά στη συνεργασία και στην ανταλλαγή πληροφοριών, πρώτα απ' όλα μεταξύ Ευρωπαίων, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Τρίτον, όταν ετοιμάζουμε νέες ρυθμίσεις, θα πρέπει να ξέρουμε γιατί αποθήκευση, διατήρηση δεδομένων μιλάμε. Και η διατήρηση να είναι μόνο η απαραίτητα αναγκαία και όχι παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των δικαστηρίων που είπαμε πριν. Πρέπει να υπάρχουν αρκετές ρήτρες ασφαλείας που θα έχουν ασωματωθεί στις νέες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να υπάρχει ακρίβεια, να υπάρχει αξιοπιστία και ασφάλεια στην επεξεργασία δεδομένων. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως να είναι τα βιομετρικά στοιχεία. Μόνο αν υπάρχει μια τέτοια ισορροπία μπορούμε να καταλήξουμε σε σωστές επιλογές και να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή. Εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην Ευρώπη, όταν ανταλλάσσουν πληροφορίες και δεδομένα, να ξέρουν ότι είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες που έχουν και ότι δεν θα χαθούν. Να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτούς που εκπονούν την πολιτική και τις αρχές επιβολής του νόμου διότι αυτές οι τελευταίες πρέπει να νιώθουν ότι είναι χρήσιμες. Επίσης εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτούς που εκπονούν την πολιτική και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Γιατί και τελευταίοι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Και τέλος και πιο σημαντικό, ίσως να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτούς που εκπονούν τον νόμο και τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη. Μόνο τότε νέα μέτρα θα μπορέσουν να υιοθετηθούν εφόσον είναι αναγκαία βέβαια, και να ε, είναι αποτελεσματικά για να προστατεύσουμε την ασφάλεια και να μην υπονομεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγήτρια. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία τέθηκαν, αλλά πρώτα θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο του Γερμανικού, της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, τον κύριο Όστερμαν. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να είναι διαφορετικό ο κύριο στόχο των ευφυών συνόρων, αλλά πρέπει να παραγνωρίζουμε και τη σημασία τη ασφάλεια, τη ασφάλειας. ασφάλεια. Το να γνωρίζουμε δηλαδή το πού και πότε κάποιο έχει περάσει τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να δώσει πολύ σημαντικέ πληροφορίε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αποτροπή των τρομοκρατικών υποθέσεων, αλλά και για την ε, καταπολέμηση τη υπερσυνοριακή εγκληματικότητα, όπω άλλωστε ο κύριο Σελάν μα εξέθεσε ήδη. Περιμένετε δύο λεπτάκια να βεβαιωθούμε ότι είναι αναμένα όλα τα μικρόφωνα. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξασφαλιστεί πρόσβαση για τις αρχές ασφαλείας. Θα ήταν μέγα σφάλμα να μην διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές, να είναι αποκομμένες από τις σημαντικές αυτές πληροφορίες οι αρχές ασφαλείας και νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις οι οποίες και θα εξασφαλίζουν απαντήσεις για την ασφάλεια αλλά και θα πληρούν τις ε, προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συστήσαμε και χτες. Για μένα και δεδομένου ότι είναι τόσο σημαντικό ο κίνδυνο τρομοκρατική απειλή, ερώτημα δεν πρέπει να είναι το εάν θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για τι αρχέ ασφαλεία και επιβολή του νόμου, αλλά το πώ θα έχουν πρόσβαση αρχέ ασφαλεία και ε, επιβολή του νόμου. Πρέπει να γίνεται λοιπόν κατά τρόπο απρόσκοπτο και χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, με μια ταχεία αξιολόγηση για να εξοικονομήσουμε και σε κόστος. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, ο κύριος Σεμπαστιάν Κουντζάλης από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Μαγκαλάης. Θα ήθελα καταρχάς να αξιολογήσω πάρα πολύ θετικά την πραγματοβουλία αυτή για την συγκεκριμένη συνάντηση για το πακέτο για τα εφή σύνορα. Είναι βασικό να μαθαίνει κανείς από τις εμπειρίες και από τις πληροφορίες τις οποίες έδωσαν σήμερα αλλά και χτες γύρω από τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να θέσω. Καταρχάς ένα γενικό θέμα σχετικά με την κυβέρνηση της Ισπανίας και τη θέση της Ισπανίας μάλλον γύρω από, το, την προτινόμενη νομοθετική ρύθμιση. Θα ήθελα να πω ότι η Ισπανική Βουλή είχε ήδη την δυνατότητα να συζητήσει τις νομοθετικές προτάσεις τις οποίες παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ισπανική Βουλή θα εγκρίνει την εισαγωγή ενός συστήματος ελέγχου εισόδων-εξόδων που θα διευκολύνει τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων γύρω από θέματα όπως η μετανάστευση. Ε, και γι' αυτό επιδιώκουμε την βελτίωση της διαχείρισης μέσω και του ε, Μητρώου Καταγεγραμμένων Ταξιδιωτών. Τώρα για τις αστυνομικές αρχές είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι αστυνομικές αρχές ε, τα συστήματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Ο κύριος Σελένα μας έδωσε μια σωστή και αναλυτική παρουσίαση των κινδύνων τις οποίους αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι το θέμα τίθεται αυτή τη στιγμή ε, ε, έχει λειτουργήσει εδώ και δύο χρόνια και έχει αξιολογηθεί σαν θετική ή παρούσα ε, νομοθετική πρόταση. Οι παρεμβάσεις των συναδέλφων χτες και σήμερα έδειξαν ότι υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες για την πρόσβαση των αστυνομικών αρχών εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες και να αναφερθώ στις λεπτομέρειες αυτές. Είναι όμως κάτι το οποίο πράγματι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η πρόσβαση των αστυνομικών αρχών δεν μπορεί να είναι απεριόριστη και άκρητη και να φύγει τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως είπε η κυρία Μπράουερ απαιτείται μια ολόκληρη σειρά εγγυήσεων για να διασφαλιστεί η ισορροπία. Ο κύριος Διαστεμέρα ε, σημείωσε τα θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και είπε τις αμφιβολίες οι οποίες ε, ε, αναφέρθηκε στις αμφιβολίες οι οποίες γεννούνται. Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι όλοι Είμαστε ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της τρομοκρατίας και αναζητούμε τις ρίζες των τρομοκρατικών επιθέσεων και αναζητούμε κάθε δυνατό τρόπο καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να διευκολύνουμε ε, την προσπάθεια αυτή και θα πρέπει να υπάρχει επαρκής περίοδος διατήρησης των στοιχείων για να αποφεύγουμε επαναληπτικές καταγραφές και μητρώα ε, τα οποία θα επιτρέπουν βέβαια ε, την ε, έρευνα κάποιων φαινομένων. Να αναφερθώ σε αυτό στο οποίο κατέληξε η κυρία Μπράουερ. Απαιτείται εμπιστοσύνη, απαιτείται η εγγύηση για ελευθερία και ασφάλεια. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ρεβόντα Λόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η φιλοδοξία του πακέτου αυτού είναι διπλή, να διευκολύνει την κινητικότητα για τους πολίτες τρίτων χωρών που ε, ταξιδεύουν συχνά και δεύτερον να διευκολύνει τις δυνατότητες περάσματος των εξωτερικών συνόρων. Ε, τίθεται εδώ και το θέμα της χρήσης από πλευράς των αστυνομικών αρχών στα στοιχεία ε, τα ε, σύνοριακά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν επιπλοκές για το FES σύστημα ελέγχου σύνορων. Σημαίνει ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους καταπολεμούμε φαινόμενα όπως η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η πρόσβαση από πλευρά των αστυνομικών αρχών θα πρέπει να είναι πλαισιωμένη από τις ανάγκες, την αναλογικότητα και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δοθούν εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε άραγε συγκεκριμένα στοιχεία για το κατά πόσον βάσεις δεδομένων όπως το VIS και το SIS βοηθούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα λίγο περισσότερα στοιχεία. Και η διευκόλυνση περάσματος στα σύνορα θα βελτιώσει την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν όλα αυτά να είναι συμβατοί στόχοι στο εσωτερικό ενός ενιαίου συστήματος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο από τη Λιθουανία. Σετ Μπάρς. να e, Ευχαριστώ πολύ, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που υποστήριξαν τη δυνατότητα για πρόσβαση στις ε, αρχές ασφαλείας για τα συστήματα εισόδων-εξόδων. Εμείς από τη Λιθουανία βλέπουμε τη μεγάλη σημασία της πρόσβασης αυτής. Έχουμε εθνικό σύστημα εισόδων-εξόδων και μπορώ να σας εξηγήσω από την εμπειρία μας πόσο χρήσιμη είναι η αξιοποίησή του για τις αστυνομικές και τις τελωνιακές αρχές ε, τόσο στην διαλεύκανση όσο και στην αποτροπή εγκλημάτων. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις χώρες εκείνες και τις ε, αρχές οι οποίες τοποθετούνται υπέρ της προσβάσεως για τις αρχές της, της τάξης και του νόμου στα δεδομένα αυτά. Υπάρχουν πολλές χώρες που τοποθετήθηκαν υπέρ, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ελβετία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα μετατραπεί η πρόσβαση αυτή σε πρωταρχικό στόχο του συστήματος συν Όχι, πρέπει να παραμένει πάντα δευτερεύον παρεμπίπτων ε, στόχος. Επίσης πρέπει να συστήσουμε το κόστος της επενδύσεως και το τι θα κερδίσουμε από μια τέτοια επένδυση. Η πρόσβαση στα δεδομένα θα συμβάλλει ασφαλώς. Ο κύριος Διέσδε Μέρα μιλάει για την προστασία των δεδομένων, για τη σημασία της ψυχής αυτής. Η επιθεώρηση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Λιθουανίας έχει ε, γνωμοδοτήσει, έχει αποστείλει τη γνωμοδότηση της στην αντίστοιχη Επιτροπή του Λιθουανικού Κοινοβουλίου και η γνωμοδότηση αυτή κατηγορηματικά τοποθετούνταν στις θέσεις της ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Δίας Δεμέρα μας είπε ότι μπορεί να χρησιμοποιούν διάφορες αστυνομικέ αρχές την, ε, την πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, αστυνομία, χωροφυλακή, στρατοχωροφυλακή κτλ. Εμείς έχουμε ένα ιδιάζον σύστημα που αντιστοιχεί πιστεύω στη στράτο στη Λιθουανία. Ε, πάντως το σημαντικό δεν είναι αυτό οι αρχές που έχουν πρόσβαση όσο οι κανόνες με βάση τους οποίους θα εξασφαλίσετε αυτή η πρόσβαση και η τήρησή τους. Κύριος στόχος είναι ο προσδιορισμός της κλίμακας εκείνων των στοιχείων που θα διαβιβάζονται και ασφαλώς θα πρέπει να τηρείται πάντα η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που μας παρουσιάστηκε σήμερα. Εμείς βλέπουμε ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται κατά το ταχύτερο δυνατό διάστημα. Αμέσως δηλαδή, αντίθετα από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να είναι ανοιχτή στις αρχές της, του νόμου και της τάξης από την πρώτη μέρα που είναι διαθέσιμες στο σύστημα. Αυτό νομίζω μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα με τα παραδείγματα των επιθέσεων στο Παρίσι και άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσωπος από τη Μάλτα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καθώς φτάνουμε προς το τέλος των εργασιών μας και συζητούμε το θέμα των εφιών ολοκληρωμένων συστημάτων για τα σύνορά μας, αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο μας εξήγησε ο κύριος Σελέν σήμερα το πρωί, δηλαδή τις Χρυσή τομή ή τη σωστή ισορροπία. Την ισορροπία όμω μπορούμε να το δούμε από πολλέ προοπτικέ. Και με βάση τι συζητήσει που ξεκίνησαν εχθέ και την έμφαση που δώσαμε στην ανάγκη για νέα συστήματα που θα διευκολύνουν τη διέλευση των συνόρων, που θα καθιστούν ευχερέστερη ε, την διέλευση και με αυξημένες ροές επιβατών που θέλουν να περάσουν τα ε, ευρωπαϊκά σύνορα. Φτάνουμε τώρα στο τέλος της συναντησής μας να συζητήσουμε τη χρήση των ίδιων αυτών εργαλείων για την ενίσχυση της ασφάλειας και της διάγνωσης προβλημάτων ή κινδύνων προς την ασφάλεια. Κάποιος είχε νωρίτερα ερωτήσει αν πρόκειται για συμβατούς στόχους. Εγώ νομίζω ότι η χρυσή, ε, χρυσή τομή, η άριστη ισορροπία είναι ακριβώς αυτό, το να καταστήσουμε συμβατούς τους στόχους. Τα ε, ίδια ηλεκτρονικά στοιχεία που θα διευκολύνουν τη διέλευση των συνόρων θα είναι και τα στοιχεία τα οποία θα μας ε, δίνουν δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας. Για την ισορροπία όμως θα πρέπει πιστεύω να υποδείξουμε και μια άλλη οπτική γωνία. Δηλαδή εξισορρόπηση μεταξύ των μέτρων που χρειάζονται και ώστε δυνατόν ελαχιστοποίηση των μέτρων αυτών προκειμένου να μην παραβιάζονται ή να μην υπάρχει κίνδυνο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ήδη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που τονίζει του όρου αποτελεσματικότητα και αναλογικότητα. Αναλογικότητα συνεπάγεται ε, ελάχιστη ντεμίνιμης προσέγγιση, όσο λιγότερα δεδομένα τόσο λιγότερα ε, αναγκαία, είναι αναγκαία, τόσο λιγότερο θα διατίθενται. Όσο λιγότερη η ανάγκη για διακράτηση δεδομένων, τόσο μικρότερο και το διάστημα διακράτησής τους. Επίσης, αναφέρθηκε ο όρος μοσαϊκό. Έχουμε πολλές πληροφορίες κατακαιρματισμένες, πολλά κομμάτια πληροφοριών, πολλά στοιχεία από τα συστήματά μας, όπως το σύστημα ε, ενημέρου πληροφοριών, βατήριων και ούτω καθεξής. Που όμως πρέπει να ρωτήσουμε, τα χρησιμοποιούμε ήδη αυτή τη στιγμή όπως χρειάζεται. Αλλά έστω ότι προχωρούμε στο, μοσαϊκό αυτό, θα είναι επαρκές το σύστημα για να ενώνει τα κομμάτια και να ανοίγει μια καθαρή εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν η ιδέα του πάζλι, του μοσαϊκού, για μένα έχει μεγάλη σημασία. Και υπό το φως των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων που είδαμε στην Ευρώπη πρόσφατα, ότι δηλαδή πολύ συχνά το ζήτημα δεν ήταν ότι δεν είχαμε διαθέσιμες πληροφορίες για άτομα που είχαν μάλιστα αναγνωριστεί και εντοπιστεί, αλλά τώρα αναγνωριζόταν ως αντίστοιχο το επίπεδο κινδύνου των συστημάτων που αναγνωρίζουν τα συστήματα ή αν είχε υποβαθμιστεί από κάποιο σύστημα ο κίνδυνος, δηλαδή αν επικοινωνούν μεταξύ του τα συστήματα. Και έτσι φτάνουμε σε μια ευρύτερη διαθεσιμότητα των διαφορετικών κομματιών στοιχείων. Όταν την έχουμε αυτήν, τότε πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα, το δυναμικό, τα μέτρα που εξασφαλίζουν το δυναμικό και εξασφαλίζουν την συμπίληση και την ενοποίηση σε ένα ε, σώμα λειτουργικό των στοιχείων αυτών. Εγώ προερχομένως από τη Μάλτα βλέπω και μια άλλη πτυχή του προβλήματος, τις πολύ μεγάλες ροές των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στη χώρα μου. Ενώ ταυτόχρονα θέλω και να υποστηρίξω και να ενισχύσω τον τακτό και ομαλό, τον καλό τουρισμό που θα έρχεται με αυξημένες ροές. Αυτό νομίζω θα πρέπει να απαντηθεί σαν ένα ερώτημα το οποίο δίνει και την κατακλείδα των εργασιών μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντυπρέ, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ντεπρέ, λέγομαι. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές για την ποιότητα των παρουσιάσεών του σήμερα το πρωί. Πολύ καλές. Να ρωτήσω κάτι την κύριε Μπράουερ πρώτα απ' όλα. Ομολογώ ότι ένιωσα κάπως περίεργα όταν σας άκουσα να μιλάτε για τη συνεργασία. Ρωτάω λοιπόν, από πλευράς προστασίας του ιδιωτικού βίου, έλεγχος δεδομένων κτλ. Δεν είσαστε πιο πολύ υπέρ των εθνικών συστημάτων και της συνεργασίας μεταξύ εθνικών συστημάτων παρά υπέρ ενός ευρωπαϊκού συστήματος. Ένιωσα ότι η καρδιά σας ήταν πιο πολύ στο πρώτο. Αν δεν είναι έτσι, τότε ερμήνευσα στραβά αυτά που είπατε. Δεύτερον, όσον αφορά την αναγκαιότητα. Όταν πρόκειται για την εφαρμογή ενός συστήματος και την αναλογικότητα. Είναι αλήθεια ότι η απόφαση λέει ότι πρέπει να παίρνουμε χ δεδομένα για να καλύψουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, αλλά να μην είναι δυσανάλογο. Αν όμως το συνδυάσετε με μια άλλη πηγή, φυσικά και πρέπει να είσαστε επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένου ανθρώπου. Και αν είσαστε επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένου ανθρώπου, του τζιχαντιστέ για παράδειγμα, έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Χρώμα και άλλα χαρακτηριστικά. Ε, θα σας πούνε ε, ρατσιστή. Αν λοιπόν αμφισβητείτε τη δυνατότητα να πάρετε γενικές πληροφορίες από διάφορους που δεν θα χρησιμοποιήσετε παρά μόνο αν συνδυαζόμενες με κάποιες άλλες πηγές σας κάνουν να πιστέψετε ότι πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε. Αυτό δηλαδή που εσείς καταγγέλλετε δεν αντικαθίσταται τελικά με κάτι χειρότερο. που συνδυάζεται με χώρες ή με περιπτώσεις πιο προβληματικές. Για τον ε, κύριο Σελέ. Κοιτάξτε, ναι, πολύ μου άρεσαν αυτά που είπατε. Όπως είπε και ο Μαλτέζος συνάδελφος, μας έπεισαν προς το παρόν για διάφορα συστήματα όπως και εκείνο εισόδων-εξόδων. Τελικά είναι η ασφάλεια που έχει το πρώτο χέρι, ενώ στην πραγματικότητα το σύστημα αυτό το θέλαμε για να ελέγξουμε τη μετανάστευση. Αν κάποιοι έχουν μείνει υπερβολικά πολύ στην επικράτειά μας, να ξέρουμε ότι αυτό έχει συμβεί και να μπορούμε να τους βρούμε. Το πρόβλημά με το σύστημα αυτό εισόδων-εξόδων έχει να κάνει με τη συνοχή, γιατί φοβάμαι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε φοβερές δυσκολίες στο μέλλον. Οι τσιχαντιστές και πάλι, νέοι, από εμά, οι οποίοι πήγανε στο Ιράκ, στη Συρία και αλλού να πολεμήσουν, έχουν τη δικιά μας την υπηκότητα των χωρών μας. Γερμανοί, Γάλλοι, Δάνοι, Δανοί, Βέλγοι, οτιδήποτε. Το σύστημα εισόδων-εξόδων τι θα κάνει. Θα εντοπίσει τους υπηκόους τρίτων χωρών. Και όταν οι τζιχαντιστές θα επιστρέψουν, πώς θα ξέρετε ότι επέστρεψαν. Θα το ξέρετε μόνο αν έχουμε ένα ευρωπαϊκό PNR μεθαύριο. Γιατί όσοι επιστρέψουν με αεροπλάνο θα έχουν καταχωρηθεί, όπως και οι Ευρωπαίοι. Αλλά όσοι θα έρθουν οδικός, ε, τα κτλ. Δεν θα τους εντοπίσετε. Οπότε ποια είναι η συνοχή του συστήματος που θέλουμε να φτιάξουμε. Ουσιαστικά μετατοπίζουμε το πρόβλημα. Μόνο αν έρθουν με αεροπλάνο θα τους εντοπίσετε. Με το σημερινό σύστημα και σε σχέση με ό,τι λένε οι ειδικοί, ποια είναι η κύρια απειλή για τα επόμενα χρόνια, το σύστημα αυτό δεν θα εξυπηρετήσει τίποτα. Και είναι κρίμα ένα σύστημα το οποίο θα στοιχήσει τόσο ακριβά να μην δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Και ποιο θα το χρησιμοποιήσει. Αν έχουμε ένα PNR μεθαύριο ευρωπαϊκό, δεν θα χρησιμοποιείται. Άρα μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε γενικά τους μηχανισμούς και τα μέσα που έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα. Γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχει μια σαφής έλλειψη συνοχής εδώ και σοβαρά κενά. Ευχαριστούμε. Ναι, η φιλοδοξία μας είναι το τέλειο σύστημα, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, το λόγο έχει ο Σλοβανός συνάδελφος. Ή συνάδελφος, Ηλιάνα Κόζοβιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση αυτή και είναι χρήσιμο για όλους το να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε. Να πω ότι η Σλοβενία θεωρεί ότι είναι θετικά τα μέτρα τα οποία προτείνονται στον τομέα των εφιών συνόρων. Έχουμε όμως και ορισμένες επιφυλάξεις. Μία από αυτές είναι το θέμα της οικονομικής επιβάρυνσης και το άλλο είναι το θέμα της διαλειτουργικότητας. Αλλά αυτό που μας απασχολεί ιδιαιτέρως είναι τα θέματα που τίθενται από τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με λανθασμένο τρόπο και αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για όλους. Το σύστημα αυτό λοιπόν αν χρησιμοποιηθεί λάθος ε, δεν θα εξυπηρετήσει τον στόχο τον οποίο αναζητούμε. Η ασφάλεια είναι μία από τις πιο βασικές αξίες ε, τις οποίες επιδιώκουμε. Έχουμε ζήσει πολλά χρόνια ε, εν ειρήνη και τώρα η Ευρώπη φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερος πλέον ελκυστική λόγω του επίπεδου προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων και λόγω των κοινωνικών μορφών κάλυψης των αναγκών των πολιτών. Όπως είπε ο κύριος Έλεν, ένα μέτρο ή μία πρόταση δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες όταν είχαμε συναντηθεί στη συνδιάσκεψη της Ρώμης, είχαμε συζητήσει το θέμα της μετανάστευσης. και εμείς ε, είχαμε πει ότι μπορούμε να ε, εξυπηρετήσουμε με κάποιο τρόπο ικανοποιητικό τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζει η νόμιμη μετανάστευση και η ε, ε, εκτός ε, νομικού πλαισίου μετανάστευση. Γιατί η Ευρώπη είναι, ένα, μια ήπειρος που γυράσκει και γι' αυτό απαιτείται εναρμόνιση των εθνικών μας πολιτικών. Και υπάρχει επίσης και το θέμα του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας είναι η διαπολιτισμική διάσταση. Έχουμε κόσμο που έρχεται στην Ευρώπη από διαφορετικούς πολιτισμούς. Ε, μιλάμε επίσης για το θέμα της προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων Δεν ξέρω ποια είναι η τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά τα κριτήρια στα οποία αναφέρθηκε το δικαστήριο ε, παρέχει δυνατότητες ανάγνωσης ε, της κατάστασης. Επόμενος ομιλητής. Ο Ιγνάσιο Κασία από την Ελβετία. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ γιατί προσεκάλεσε και την Ελβετική Αντιπροσωπεία, αν και η Ελβετία ε, δεν συμμετέχει άμεσα στις διαδικασίες Σέγγεν. Παρ' όλα αυτά η χώρα μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για τα θέματα αυτά του πακέτου των ευφυών συνόρων. έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Μπράουερ, καθηγήτρια Μπράουερ, για την ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ευρωπόλ. Δεν έχω βρει όμως στα έγγραφα στα οποία μας έχουν αποσταλεί μέχρι τώρα κάποιες αναφορές για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να κατανοήσω καλύτερα τι είδους μορφή συνεργασία και τι διευκρινήσεις μπορούν να δοθούν πριν προχωρήσουμε στο σχέδιο Smart Borders. Δεύτερον, όλοι στα κοινοβούλια μας έχουμε βιώσει τις εμπειρίες της δυσκολίας των μεγάλων πληροφορικών συστημάτων με τεράστιο κόστος και έχουμε δει και αποτυχίες τεχνικές και τεχνολογικές. Το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θέτω με πολιτικό τρόπο και το θέτω και σε άλλα κοινοβούλια. Θα ήθελα να μάθω τι είναι τελικά πιο σημαντικό σε πολιτικό επίπεδο. Η ασφάλεια των εξωτερικών σύνορων. Σε έναν κόσμο ανασφαλή λόγω όλων αυτών των τρομοκρατικών ε, ε, ενεργειών ή είναι πιο σημαντικό να διευκολύνει κανείς και να επιταχύνει ε, τις διαδικασίες στα εξωτερικά. Το αυγό του Κολόμβου θα ήταν φυσικά να συνδυάσει τις δύο αυτές διαδικασίες. Ο κύριος Διασταλμέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λόγια για να αντιδράσω σε κάποια σχόλια που ακούσαμε. Χωρίς βέβαια να θέλω να πω ότι εγώ ξέρω. Λέμε κάποια πράγματα από ένστικτο ή θεωρητικά. Εντάξει, απόλυτα θεμητό. Και υπάρχουν και άλλες παραβάσεις όπως αυτή που έχει να κάνει με την εμπειρία, με τη γνώση δηλαδή της πραγματικότητας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω κάποια πράγματα χωρίς να θέλω να διορθώσω τους προλαλήσαντες, αλλά για να σας πω ποια είναι η δικιά μου θέση, η θέση δηλαδή του εισηγητή για αυτά τα θέματα. Χτες μίλησα για το πρωτογενές δικαίωμα, το πρωταρχικό, που έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα. Άρθρο 8 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα λέει όλα. Άρθρο 16 της Εθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάλι θεμελία δικαιώματα, προστασία τους. Δηλαδή, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αδιέρετα. Είναι σημαντικό και το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο και το δικαίωμα στην ασφάλεια. Αναμφίβολα. Δεύτερον, συμφωνώ με κάποιους συναδέρφους βέβαια. Ακούσαμε για την εμπιστοσύνη. Πρέπει να θέλουμε να κάνουμε. Ναι, αλλά την εμπιστοσύνη μπορεί κανείς να την ορίσει, αλλά το βασικό είναι να την νιώσει. Κατά τη γνώμη μου, αδίκως ακούσαμε ότι η Europol δεν λειτουργεί καλά. Εγώ θα σας πω ναι. Ήμουνα μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, κυρία μου, και ήμουνα και συγητής εκεί και είμαι ο εισηγητής του κανονισμού για τη Europol. Και σας λέω ότι ναι, λειτουργεί. Ωραία. Επιδέχεται βελτιώσεις, ε, τελειοποίηση, ναι. Λειτουργεί όμως. Το PNR είναι ένα επιπλέον εργαλείο. Και όταν λέμε ότι θα μπορούσε να παραβιάσει το χώρο του ιδιωτικού βίου, διαβάστε την νομοθετική πρόταση, η οποία προστατεύει τον ιδιωτικό βίο και απαγορεύει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την προέλευση, τη θρησκεία, το φύλλο κλπ. Είναι νομοθετική πρόταση και αύριο ο Πύρκο θα μας παρουσιάσει τη σχετική τροποποίηση. Και υπάρχει δικαίωμα στη διόρθωση, στην πρόσβαση Πρέπει να μιλάμε με επιχειρήματα, θεωρητικά, ναι, αλλά και βάσει της εμπειρίας μας. Και για να ολοκληρώσω, πολλά θα είχα να σας πω. Κοιτάξτε, όταν μιλάς κάθε φορά σε ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα, αλλά προσέχω τι λες. Πολύ. Την προηγούμενη φορά από, μάλλον πριν από λίγο, από τις κάτω χώρες, ακούσαμε τι είχαν να μας πούνε και μετά ακούσαμε τη Γερμανία και τη Μάλτα. Όλα αυτά τι σημαίνουν, διαλειτουργικότητα μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας. Αλλά δεν είναι το μόνο, υπάρχουν και άλλα μέσα. Αν αυτά τα άλλα, στα οποία δεν θα αναφερθώ εγώ, έχουν αναφερθεί οι άλλοι, συνεργαστούν Υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ τους δηλαδή, τι πετυχαίνουμε. Καλύτερο και πιο ευέλικτο και γρήγορο έλεγχο στα σύνορα και πετυχαίνουμε επίσης και καλύτερη προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων. Θα σταματήσω εδώ, γιατί δεν θέλω κι εγώ να καταχραστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα προσθέσω περίπλοκα ζητήματα όπως η στρατηγική πρόληψη που είναι και το πιο επίκαιρο ζήτημα. Και δίνω το λόγο στο τελευταίο μιλητή, τουλάχιστον στο δικό μου κατάλογο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να, να στήσει το λόγο. Η κυρία Άννα έχει έχετε το λόγο, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ. Έχω εργαστεί εδώ στο Κοινοβούλιο και επεξεργαστεί στρατηγικές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από την Επιτροπή, υποεπιτροπή μάλλον της Άμυνας και της Ασφάλειας. Δεν έχω αμφιβολία λοιπόν ότι η ε, διάθεση πληροφοριών και η διαλειτουργικότητα έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα εξισορροπηθεί αυτή με τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία σημειώνουν είναι σημαντικά. Όχι και είναι δικαιώματα όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά για τους πάντες αυτό ορίζει και η νομολογία του δικαστηρίου. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι είδους ισορροπία χρειάζεται για την προστασία των δεδομένων έναντι όλων. Και πιστεύω ότι η ενίσχυση της Europol και η πρόσβαση σε αυτήν του σχετικού δυναμικού των σχετικών δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντική γιατί η Europol μπορεί να διαδραματίσει ρόλο κρίσιμο και να συνεχίσει και στο μέλλον ακόμη περισσότερο κρίσιμο ρόλο να διαδραματίζει. Το ότι δεν τα καταφέρνει πάντα οφείλεται στα κράτη-μέλη γιατί εκεί εντοπίζεται η απουσία της διαλειτουργικότητας και η απουσία εμπιστοσύνης. Επί παραδείγματι σε χώρες όπως η δική μου και η δική σου, πρόεδρε, Πορτογαλία δηλαδή, όπου επί παραδείγματι δεν έχουν οι αρχές των πληροφοριών να καταγράψουν, να συλλάβουν, να ανοιχνεύσουν με νόμιμο τρόπο ε, κάποια φορά τρομοκράτες, αλλά παρόλα αυτό το πράττουν. Άρα χάνεται η εμπιστοσύνη και χάνεται και η εμπιστοσύνη μεταξύ αρχών ε, συλλογής πληροφοριών και επικοινωνία διαβίβαση των στοιχείων αυτών από τη μια χώρα στην άλλη. Άρα είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και χρειάζεται μια συνεπής προσέγγιση. Εν προκειμένου ερωτώ λοιπόν και τη γερμανική αστυνομία, μια και έχουμε γερμανική ε, Ευρώπη, Ας ρωτήσουμε για τη γερμανική αστυνομία. Για τεφή σύνορα, ερώτηση που έκανα και χθε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε μέχρι τώρα τη στακτική στάση, αλλά πάντως η εκπροσωπή πώς χθε εχθές υπεγράμμισε το πρόβλημα. Πώς λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε τα σύνορα όταν τα ανοίγουμε μόνο για αυτούς που, τους πλούσιους που μπορούν να έρθουν με τη χρυσή λεγόμενη θεώρηση και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτούς οι οποίοι μπορεί να οργανώνονται, να παραμένουν σε αδράνεια για ένα διάστημα. Είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν δυσκολίες και αντιφάσεις ως προς τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος των τσιχατιστών, των παράτυπων μεταναστών και από την άλλη θέλουμε να προωθήσουμε τον τουρισμό. Πολύ καλά, αλλά η θαγένεια οι άδειε παρανομής που χορηγούν ορισμένες χώρες της Ευρώπης σε επικούς τριτών κρατών χωρίς καμία επαλήθευση, χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν έχει σημασία αυτό το ζήτημα και για τη Γερμανία. Και βέβαια και τα άλλα ερωτήματα που πως χθες στο οποία έδωσε απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω το γεγονός ότι κανείς δεν συζητάει την εφαρμογή εφιών ελέγχων σε επιβάτες ιδιωτικών, μη στρατιωτικών αεροσκαφών ή θαλαμιγών ή σκαφών. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, μας έχουν μείνει περίπου τα 10-15 λεπτά πριν κλείσουμε και προτείνω το εξής να περιορίσουμε το χρόνο απαντήσεων για τους ομιλητές μας, 5 λεπτά ο καθένας, ώστε να τους θέσουμε και ενώπιον της τεράστιας πρόκλησης να απαντήσουν στο πολύ ευρύ αυτό φάσμα ερωτήσεων που πόθη και Θέλετε να ανταλλάξετε σειρά ή η καθηγήτρια Ντεμπράουερ λοιπόν. Εσείς έχετε το λόγο. Thank you for all. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα ξεκινήσω με κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Ίσως είπατε να υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στα ε, στους στόχους της προσπάθειας διευκόλυνσης της εισόδου και από την άλλη στα θέματα ασφαλείας. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα δύο. Έχουμε κάποια μέτρα τα οποία προτείνονται και τα οποία εφόσον εφαρμοστούν σωστά ε, δεν θα παρουσιάσουν τρομερά προβλήματα. Ίσως όμως να υπάρξουν κάποιες μικρές αντιφάσεις λόγω της ανυπαρξίας ε, ε, κάποιων κοινών κριτηρίων στην εφαρμογή των μέτρων αυτών. Είπατε ότι λόγω των διαφορών αυτών θα πρέπει εκ των προτέρων να κάνουμε κάποιες επιλογές, να προσπαθήσουμε να δούμε τι χρειαζόμαστε περισσότερο σαν βασικό στόχο τον στόχο της ε, διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ή τον στόχο της αύξησης του επίπεδου ασφαλείας. Εγώ είπα ότι στις προτάσεις οι οποίες γίνονται περιλαμβάνονται στοιχεία τα οποία τίνουν στην ε, κράτηση των συγκεκριμένων ατομικών στοιχείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εδώ θα έλεγα ότι πράγματι οι επιβάτες θα ήθελαν να υπάρχει μια ε, τακτοποίηση στα Μητρώα η οποία να μην οδηγεί στην κράτηση των στοιχείων που περιλαμβάνουν για υπερβολικά μεγάλη ε, χρονική περίοδο. Κατανοώ τις ανησυχίες και σέβομαι τις ανησυχίες αυτές. Ταυτόχρονα εγώ εκτιμώ την προσπάθεια την οποία κάνουν οι εσωτερικές ε, δυνάμεις ασφαλείας, οι υπηρεσίες γενικότερα που ασχολούνται με τα θέματα ασφαλείας ε, και κατανοώ και τους λόγους που τους οδηγούν να ζητούν μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης των στοιχείων αυτών. Το θέμα είναι να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Τώρα, για το πρόγραμμα αυτό ε, για τις ε, θεωρήσεις για τους ταξιδιώτες. Θα πρέπει κανείς να είναι βέβαιος για τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται και τα οποία πρέπει να τηρούνται για να εντάσσεται κάποιος επιβάτης σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε ότι βασικός στόχος είναι ο έλεγχος της κινητικότητας με την έννοια της διευκόλυνσης της κινητικότητας. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραβλέψουμε τα προβλήματα ασφαλείας. Μία παρατήρηση τώρα μετά από αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του Λιθουανικού Κοινοβουλίου ε, για την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά των αστυνομικών αρχών. Πράγματι κάθε οργάνωση η οποία αποδεικνύει, οργάνωση εννοώ τήρησης τάξης, ασφάλειας κτλ, η οποία αποδεικνύει ότι έχει ανάγκη ε, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Και εδώ θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία και τι πρόσβαση έχουν οι αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες. Πάντως δεν μπορεί να υπάρχει άκρητη ανεξέλεγκτη χρήση, θα πρέπει να τεκμηριώνεται το αίτημα για την χρήση των στοιχείων αυτών κατά περίπτωση. Δεν μιλάμε για μια γενίκευση των στοιχείων αυτών. Απαιτείται δικαστικός επίσης έλεγχος, κάτι το οποίο βέβαια κατά περίπτωση μπορεί να παίρνει διαφορετική μορφή. Για τον κύριο Ντεπρέ κατανόησε ε, σωστά αυτό που είπα για τη διατήρηση ε, του εθνικού συστήματος, αλλά εγώ εννοούσα ίσως κάτι το διαφορετικό. Εγώ εννοούσα ότι πράγματι από τα στοιχεία τα οποία έχουν στην διάθεσή τους οι εθνικές αρχές μπορούν να ωφεληθούν όταν λειτουργήσει το νέο σύστημα και εκεί θα τεθεί το θέμα της ε, κατανομής ε, των στοιχείων που άπτονται θεμάτων όπως η εσωτερική ασφάλεια στα κράτη-μέλη. Ε, εκεί πράγματι η σωστή κυκλοφορία των πληροφοριών και η ενημέρωση μπορεί να είναι πολύτιμη. Μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και μπορεί να βοηθήσει και ενδιάμεσες υπηρεσίες όπως η Ευρωπόλου. για το θέμα της αναλογικότητας. Και για το θέμα που έθεσε η Σλοβένα ε, εκπρόσωπος, να πω εδώ ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, προφανώς ε, δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια. Δηλαδή πολλές φορές ο σεβασμός των προσωπικών δικαιωμάτων βοηθά ε, την διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας μιας χώρας. Είναι σαφές λοιπόν ότι η χρήση των στοιχείων αυτών και η δυνατότητα ε, χρησιμοποίησης ακριβώς αυτών των στοιχείων είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο κατά περίπτωση. Αυτά νομίζω ότι έδωσα τις περισσότερες ε, απαντήσεις που μου ζητήθηκαν. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η σειρά σας κύριε Σελέν. θα είναι μεγάλη πρόκληση. Να δώσω απάντηση με βάση τη δουλειά μου στην καταπολέμηση της δημοκρατίας και του εγκλήματος στις ερωτήσεις αλλά θα προσπαθήσω. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα για την αναλογικότητα. Ε, ουσιαστικά πρόκειται για πολύ λιγότερα πρόσωπα που προσπαθούμε να ε, διαγνώσουμε. Όμως, όμως πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, θέλω να το λάβετε αυτό υπόψη, μπορούν να κάνουν τεράστια ζημιά στην Ευρώπη. Και εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε θεμελιώδη δικαιώματα ανθρώπων, τα οποία θα παραβιαστούν ε, εάν ε, προκύψει τρομοκρατική επίθεση. Αυτό πρέπει να το, λάβουμε, να το λαμβάνουμε υπόψη όταν εξετάζουμε την αναλογικότητα των μέτρων. Αναφέρθηκαν διάφορα μέσα σύστημα πληροφοριών Schengen, σύστημα πληροφοριών θεώρησης διαβατηρίου, γιατί δεν αρκούν. Δεν είναι δυνατόν με ένα κατσαβίδι να ε, χτυπήσετε πρέκι, θα έλεγα. Ε, δηλαδή δεν είναι κατάλληλα τα μέσα. Πρέπει να έχουμε μια συνολική λύση, αυτό αναζητούμε, και πρέπει να ομολογήσω ξεκάθαρα ότι μέχρι τώρα έχουμε αποτύχει στο στόχο αυτό. Δεν έχουμε μπορέσει δηλαδή να αναπτύξουμε τη συνολική εικόνα ή να περιγράψουμε τις συνολικές ανάγκες που θα οδηγούσαν στην δικτύωση των στοιχείων. Εμείς ως αρχή ε, ασφάλειας είμαστε απολύτως ε, ε, συμφιλειωμένοι με την ιδέα ότι θα είμαστε δευτερεύων παράγων δευτεραγωνιστές σε αυτήν την επεξεργασία, διάθεση και παρακράτηση δεδομένων ότι ο κύριος παράγωνο, πρωταγωνιστής θα είναι οι αρχές ε, φύλαξης των συνόρων για τη μετανάστευση. Αλλά μπορούμε νομίζω και εμείς να συμμετάσχουμε. Η προστασία των δεδομένων που αναφέρθηκε, νομίζω ότι αφορά όλες τις αρχές, είτε πρόκειται για αστυνομικέ, στρατιωτικές, είτε καθαρά πολιτικού χαρακτήρα αρχές όπως αυτές που έχουν να κάνουν με την διαχείριση της μετανάστευσης. Όλες πρέπει να σέβονται τα προσωπικά δεδομένα και να αναπτύσσουν σχετικά συστήματα που θα προβλέπουν τους όρους χρήσης ανεξαρτήτως του αν έχουν καθαρά πολιτικό, δηλαδή μη στρατιωτικό ή περισσότερο στρατιωτικό χαρακτήρα οι αρχές αυτές. Από τη Γαλλία ακούστηκε το ερώτημα εάν το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και θεωρήσεων θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν. Βεβαίως και αξιοποιούνται ήδη για την καταπολόμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, το SES και το VIS είναι κέρια συστήματα. πρέπει να ξέρετε ότι έχει κεντρική σημασία, έχουν κεντρική σημασία τα συστήματα αυτά, όπως και η Europol. Έχει τεράστια σημασία. Δεν μπορούμε να την υποτιμούμε, ούτε να την υπονομεύουμε. Πρόκειται για ένα κεντρική σημασία σε εργαλείο, πρέπει να αναπτυχθεί, αλλά και δεν πρέπει και να επιβαρύνεται υπερβολικά με ε, ε, ε, καθήκοντα τα οποία δεν μπορεί να επιτελέσει. Ο έλεγχος των συνόρων ανήκει στον έλεγχο των συνόρων. Δεν μπορεί να αναλάβει τα πάντα η Europol. Πάντως είναι ένα πολύτιμο και σημαντικό εργαλείο και πρέπει να ενισχύεται. Σε σχέση με τους τζιχατιστές, με ταυτότητα ευρωπαϊκή, που πάνε στη Συρία, εκπαιδεύονται εκεί και επανέρχονται. Ναι. Μιλούμε εδώ όντω για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό είναι πάλι μέρος της πραγματικότητας, γιατί το 1 τρίτο των ατόμων αυτών είναι υπήκοοι τρίτων κρατών, τουλάχιστον στη Γερμανία, και όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει και αυτούς να τους δούμε. Δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στα τραγικά περιστατικά των τελευταίων μηνών. Υπάρχουν διαφορετικά σενάρια που θα πρέπει να αναπτυχθούν για να κοιτάξουμε προς το μέλλον στα επόμενα 5-6 χρόνια, γιατί έχουμε το homegrown terrorism, έχουμε δηλαδή την εγχώρια τρομοκρατία, όπου μόνο εθνικά μέτρα και μέτρα μπορούν να αναπτυχθούν συνεργασία με τα ε, γειτονικά κράτη μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Μετά έχουμε εκείνους οι οποίοι μεταβαίνουν σε περιοχές κρίσης και εκεί ριζοσπαστικοποιούνται, δεύτερο σενάριο, όπου μπορούμε ένα, να αξιοποιήσουμε για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού ένα πακέτο ευφυών μέτρων. Και έχουμε επίσης αυτούς τους οι οποίοι ήδη ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις ε, και αναπτύσσουν δραστηριότητα σε διάφορες ε, δραστηριότητες και επιθέσεις που μπορεί να είναι είτε υπήκοοι των κρατών μελών είτε υπήκοοι τρίτων κρατών. Εδώ εντοπίστε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μπορεί νομίζω ε, η προοπτική που συζητείτε εσείς να φέρει πολύ ε, μεγάλη βοήθεια. Η Ισλαμική Τζιχάντε, παραδείγματι, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε κάνει μια προσπάθεια για επέκταση στη Γερμανία ε, όμως, ε, και ναι, είχαμε παράγοντες που δραστηριοποιήθηκαν με ταυτότητα ευρωπαϊκή. Από την άλλη, είχαμε τις περίφημες εκείνες απειλούμενες ε, επιθέσεις κατά του, της χριστουγεννιάτικης αγοράς του Στρασβούργου από υπηκόους τρίτων κρατών που είχαν, εντα, ε, είχαν εισέλθει στη χώρα για να αναπτύξουν εκεί τρομοκρατική του δραστηριότητα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλούμε για μεμονωμένα περιστατικά και να προσπαθούμε να βρούμε με βάση μεμονωμένε καταστάσει ε, λύσει που θα καλύπτουν κάθε ενδεχόμενο, αλλά πρέπει να βρούμε ευφυεί λύσει που θα μα επιτρέψουν τη βέλτιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Ελπίζοντα ότι μπόρεσα έστω συνοπτικά να δώσω απαντήσεις στα ερωτηματικά σας ε, διατελώ στην διάθεσή σας εάν τυχόν υπάρχει κάτι συμπληρωματικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ευθύς αμέσω θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι. Θα δώσω και πάλι τα ενία στην ε, πρόεδρό μας. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασης αυτής. Θα δώσω το λόγο στους εισηγητές λοιπόν. Στην κυρία Φαγιών. Α, όχι. Πρώτο κύριος Δίαθ Δεμέρα, που πρέπει να φύγει, λέει η κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ευχαριστώ σε όλους τους συναδέρφους, τόσο από τα Εθνικά Κοινοβούλια όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας βοήθησαν πολύ με τα σχόλιά τους και σίγουρα θα συνεχίσουν να μας βοηθούν για να προχωρήσουμε με την νομοθετική αυτή δέσμη που είναι τόσο περίπλοκη. Όντω έχω κάποια ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο, γι' αυτό θα φύγω αμέσως μετά. Αλλά η Τάνια Φαγιών, έτσι καλώς πιστεύω ότι θα συνοψίσει πολύ καλύτερα τα συμπεράσματα. Πριν φύγω όμως, μόνο να σχολιάσω λίγα πράγματα και να πω κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, θα υπάρξει μια νέα νομοθετική δέσμη το 2016. Γι' αυτό χρειάζονται συζητήσεις, πολλές συζητήσεις σαν τη σημερινή, για να καθορίσουμε πώς θέλουμε, ποια μορφή θέλουμε να έχει νέα νομοθετική ρύθμιση. Δεύτερον, ποια είναι η σημερινή κατάσταση έχουμε προβλήματα στην ε, διαχείριση των διελεύσεων στα σύνορα. Κανένα σύστημα όμως δεν πρόκειται να φτάνει από μόνο του τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν τρεις χώρες που ήδη εφαρμόσουν το σύστημα εισόδων-εξόδων που δεν είναι όμως διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Πρέπει να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα και το κόστος του συστήματος. Για να διαχειριστούμε όμως αυτή την κατάσταση χρειαζόμαστε πράγματι ένα ε, ενωσιακό μέσο. Στη συνέχεια όλοι συμφωνούν για την αναγκαιότητα να ορίσουμε πιο ξεκάθαρα τους στόχους του συστήματος εισόδων και εξόδων, που είναι και το δικό μου θέμα. Από τα κράτη-μέλη οι περισσότεροι σχεδόν όλοι λένε ότι ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η διαχείριση των ταξιδιωτικών ροών και στη συνέχεια το θέμα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος που είναι θέματα των σώματων ασφαλείας. Το Κοινοβούλιο επίσης συμφωνεί με αυτό για το πιο είναι ο κύριος στόχος δηλαδή. Κάποιοι όμως βουλευτές ζητούν και πολύ σωστά να υπάρχει πρόβλεψη για αιτιολόγηση προκειμένου να μπορούν και οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά που είναι ο δευτερεύον στόχος. Για την πρόσβαση αυτή από τα Εθνικά Κοινοβούλια κατάλαβα ότι υπάρχει μεγάλη στήριξη στα όσα είπα εγώ. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει μεγαλύτερη αιτιολόγηση. πρέπει να δούμε και τι έχει αποφέρει μέχρι τώρα το σύστημα VIS. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο status quo, δεδομένου ότι αυξάνονται τα εξωτερικές ροές στα σύνορα, είναι αναγκαίο να καταλήξουμε σε ευφύς λύσεις. Το κλειδί ποιο είναι, είναι η προστασία των δεδομένων. Πρέπει να τηρούνται οι δικαστικές αποφάσεις που είναι προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς καμία αμφιβολία. Όλοι όσοι πήραν το λόγο θέλουν ένα γερό σύστημα ανταλλαγή δεδομένων. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ώστε οι πρωταρχικοί και δευτερεύοντες στόχοι να έχουν τη θέση που τους πρέπει. Όσον αφορά την χρονική διάρκεια διατήρησης των δεδομένων υπάρχει περίπου ομοφωνία ότι δεν πρέπει να συνδέεται με το κατά πόσο θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, οι αρχές επιβολής του νόμου ή όχι. Το Ουλίσε μιλάει για την διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων που εμπίπτει στις χώρες μέλη να την κάνουν, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα στη συλλογή δεδομένων κυρίως για τα βιομετρικά στοιχεία. Όσον αφορά τώρα την αρχιτεκτονική και τον προπολογισμό, η διαλειτουργικότητα ναι, να χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα συστήματα ναι, να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ό,τι έχουμε σήμερα για να μην βιαστεί πολύ ο προπολογισμό. Και τέλος, Κάρλος. Δεν πρέπει όντω να επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε με την εκτίμηση του κόστους με το σύστημα ΣΥΣ. Περιμένουμε τα τεχνικά συμπεράσματα της δοκιμαστικής περίοδου και στο μεταξύ θα συνεχίσουμε να βαθύνουμε περισσότερο στους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ από βάθος καρδίας όλους και θα τα ξαναπούμε. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Δίας μέρα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φαγιόν. Σε ευχαριστώ πολύ Κίνγκα, σας ευχαριστώ επίσης ε, και τον Αυγουστίν, Ήταν χάρα που συνεργαστήκαμε. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συμμετέχοντες για τις πολύτιμες παρεμβάσεις τους και τη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ για την οργάνωση αυτής της γραμματείας, κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο ε, για τις συζητήσεις μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν νομίζω ότι ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσες και μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε τα θέματα τα οποία σε καθημερινή βάση τίθενται στις χώρες μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τα θέματα αυτά στις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή θα προσπαθήσουμε να δούμε τα αποτελέσματα της φάσης του τεστ, του ελέγχου αυτών των προτάσεων. Θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε σωστά τα βήματα προόδου, να δούμε ακριβώς ε, τις πληροφορίες που θα μας δώσουν τα στοιχεία αυτά που θα προέλθουν από τον έλεγχο της εφαρμογής των προτάσεων περιμένοντας την επόμενη νομοθετική πρόταση το 2016. Έγιναν κάποιες παρατηρήσεις ε, ιδιαίτερα από τους ομιλητές που ζητούν να υπάρξει η προσοχή και επιφυλακτικότητα σε σχέση με την αναλογικότητα, την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή του σεβασμού ε, της πραγματικής ανάγκης από πλευράς διαφορών υπηρεσιών έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τα στοιχεία. Τίθεται επίσης από αρκετούς συναδέλφους και το θέμα του κόστους, πόσα θέλουμε να δώσουμε, πόσα θέλουμε να θυσιάσουμε για υψηλότερη ασφάλεια, ε, σε ποιο βαθμό επίσης θέλουμε να μπούμε στην ιδιωτικότητα των ταξιδιωτών και σε ποιο βαθμό θα επιτρέψουμε τέλος στις αστυνομικές αρχές να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά. Βασικός στόχος μας είναι η διευκόλυνση των πολιτών και αυτοί που χρειάζονται θεώρηση για να μπουν στον χώρο Σέγγεν συλλέγουμε ήδη ε, δακτυλοσκοπικά στοιχεία και κρατούνται αυτά τα στοιχεία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί να μην μπορέσουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το υπάρχον σύστημα, να το διευρύνουμε ίσως και γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα. Αυτά θα τεθούν στο μέλλον. Το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό βέβαια και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θυμίζω ότι εμείς ε, ήδη ε, προσπαθούμε να εργαστούμε επί τη βάση νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι μάλλον ε, ανεπαρκείς. Το έχουμε πει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη για νέα νομοθεσία. Η νέα νομοθεσία λοιπόν θα πρέπει να είναι καλύτερη και όχι να περιορίζει ακόμα περισσότερο τις ελευθερίες των πολιτών της Ένωσης και των πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες. Η πορεία μας δεν θα είναι εύκολη στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι συνεργαζόμενοι με τα κοινοβούλια των κρατών μελών θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Κυρία Φαγιόν, φτάσαμε στο τέλος της διακοινοβουλευτικής αυτής συνεδρίασης. Δεν θέλω να πω και να επαναλάβω αυτά που είπε η κυρία Φαγιόν. Σας ευχαριστώ όλες και όλους, τους ομιλητές, τους συντονιστές, τους νέους συναδέλφους που συνέβαλαν στις συζητήσεις μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα και χρήσιμα. Όπως βλέπετε, τα θέματα τα έχουν αναλάβει άξιοι εισηγητές και μπορούμε πιστεύω να προχωρήσουμε στις εργασίες μας με τρόπο καλό και υπεύθυνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Σας εύχομαι καλή επάνωδο υπενθυμίζω στους συναδέλφους της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών ότι συνεχίζουμε στις 3 το απόγευμα με την τακτική συνεδρίασή μας. Στην ίδια Ευχαριστώ.